Ja, herzlich willkommen. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε σήμερα μία έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και έχουμε σημαντικά θέματα να διεξέλθουμε στο πλαίσιο της κλιματικής προστασίας και κυρίως για το πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ελπίζω να έχετε στα χέρια σας την ημερήσια διάταξη και μπορούμε να την εγκρίνουμε όσο έχει, αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση ή παρατήρηση. Θέλετε κάτι για την ημερήσια διάταξη. Όχι. Ωραία. Εντάξει, δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα. Έχουμε όλες τις γλώσσες εκτός από τα εσθονικά και τα μαλτέζικα. Αύριο θα είναι διαφορετικά. Και αύριο έχουμε συνεδρίαση όχι σε αυτή την αίθουσα, αλλά στην αίθουσα στη 2Q2 είχαμε την ε, ακρόαση του κυρίου Μπόρκ, του υποψηφίου Επιτρόπου και φυσικά όλοι είναι προσκεκλημένοι σε αυτή την ακρόαση πέραν των μελών της Επιτροπής μας. Να κάνω λοιπόν μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα αυτό ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής αλλά και όπως έχει αποφασιστεί και εισηγητής για το θέμα αυτό και θα αναφερθώ στο θέμα της καθυστέρησης των πληστηριασμών για την εμπορία εκπομπών γνωστό ως backloading το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη νομοθετική του θητεία είχε εγκρίνει ένα πακέτο για τα θέματα ενέργειας και κλίματος, ένα συνολικό πακέτο μέτρων και δεν μπορεί να, υπάρξει, δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πακέτο σε όλη, όλο τον κόσμο. Η σπονδυλική στήλη αυτού του πακέτου και της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατεύσει το κλίμα και να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος είναι το σύστημα εμπορίας εκπομπών, ETS. Και σήμερα ακριβώς το εγχείρημα στο οποίο θέλουμε να αποδηθούμε είναι να συζητήσουμε το σύστημα αυτό εμπορίας εκπομπών. Αυτή βέβαια είναι για μένα η δεύτερη καλύτερη λύση. Η καλύτερη λύση θα ήταν μια φορολογική ρύθμιση αλλά η φορολογική ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα απαιτούσε μια ομοφωνία στο Συμβούλιο και αυτό δεν φαίνεται πολύ πιθανό. Επομένως, αυτή τη στιγμή με τις τωρινέ συγκυρίες, το σύστημα αυτό εμπορίας εκπομπών είναι η καλύτερη λύση. Βρισκόμαστε στη δεύτερη περίοδο του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Δεν μπουσουλάει πλέον, αλλά τρέχει το σύστημα αυτό. Βέβαια παρουσιάζει ακόμα και κάποιες αδυναμίες και παιδικές ασθένειες. Αλλά συγχρόνως έχουμε και τις απόρριες της οικονομικής κρίσης η οποία προέκυψε λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Και φυσικά το σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε για να λειτουργήσει προϋποθέτει μια οικονομική ανάπτυξη, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα. Και επομένως πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στο σύστημα αυτό και είναι φανερό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν, υπάρχει ένας υπερβολικός αριθμός πιστοποιητικών έναντι της ζήτησης για αυτά. 8,6 ευρώ κοστίζει ένα πιστοποιητικό σήμερα, ενώ όταν ξεκίνησε το 2008 η διαδικασία για το σύστημα αυτό, κόστιζε το κάθε πιστοποιητικό περίπου 30 ευρώ ή προβλεπόταν να κοστίζει περίπου 30 ευρώ και θεωρούσαμε ότι με μια τέτοια τιμή θα μπορούσε να παροτρύνει επενδύσεις οι οποίες θα προστάτευαν το κλίμα. Έχουμε αποφασίσει το σύστημα εμπορίας, αλλά φυσικά δεν είχαμε καθορίσει τις τιμές για, από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούσαμε φυσικά να συζητούμε και υπήρχαν διαφορετικές απόψεις για το ποια ήταν η πιο εύστοχη τιμή για τα πιστοποιητικά αυτά, αλλά δεν μπορούσαμε να το καθορίσουμε υποχρεωτικά. Αυτό θα είναι και θέμα συζήτηση με του εμπειρογνώμου. 25 Ιουλίου υπήρξε μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δική μου ερμηνεία αυτή τη πρόταση, η δική μου ανάγνωση είναι αυτή ότι θα πρέπει να υπάρξει νομική ασφάλεια σε σχέση με τα μέτρα αυτά του λεγόμενου backloading, τη μετάθεση στο χρόνο των πληστηριασμών για δικαιώματα εκπομπών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Κομισιόν να μας παρουσιάσει τα στοιχεία της πρότασης αυτής να μας ε, δείξει πώς θα πρέπει να λειτουργεί καλύτερα το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ανταποκρίθηκε στην ε, αίτησή μας η Κομισιόν. Δεν, υπάρχει, δεν είναι τώρα ιδιαίτερα μακροσκελής η πρόταση της Κομισιόν. Πρόκειται το, το θέμα της ε, έκδοσης των πιστοποιητικών και της διανομής του συζητάται σε άλλους χώρους. Αλλά αυτή τη στιγμή η Κομισιόν θέλει να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά η αγορά. Και φυσικά και για λόγους ασφάλειας δικαίου η διατύπωση της πρότασης έχει πάρει αυτήν την μορφή και φυσικά υπάρχει για, σε ορισμένους κύκλους και κάποια σύγχυση. Ορισμένοι δεν έχουν κατανοήσει ποια ακριβώς είναι η έννοια αυτής της πρότασης της Κομισιόν και υπάρχουν πολλές απορίες από την πλευρά και των μελών του Κοινοβουλίου και αντίρρηση ορισμένε φορές σε σχέση με το σύστημα της επιτροπολογίας, το οποίο συνοδεύει την λειτουργία του συστήματος. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε κάτω από πίεση χρόνου. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια πρόταση και να τύχει επεξεργασίες και έχουμε την Κόνι Χέντεγκα, την αρμόδιο επίτροπο για το περιβάλλον και έχουμε και τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, αλλά έχουμε και εκπροσώπους από τους βιομηχανικούς κλάδους, έχουμε εμπειρογνώμες που θα ακούσουμε σήμερα σε σχέση με το θέμα αυτό για τα υπέρ και τα κατά του συστήματος ETS και για το μέλλον, τη μορφή που θα πρέπει να λάβει στο μέλλον το, το σύστημα αυτό. Για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε αποφασίσει να εκπονήσουμε μια έκθεση για τα θέματα αυτά που είναι αρμόδια επί η η δική μας Επιτροπή και έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε και εγώ ο ίδιος ως συγητής να ρυθμίσουμε το χρονοδιάγραμμά μας έτσι ώστε να μπορέσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό αλλά και με την απαιτούμενη ισορροπία και σοφροσύνη για να καλύψουμε όλες τις ε, πτυχές του. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσουμε σε σχέση με τα θέματα αυτά να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα μαζί και με τις αρμόδιες επιτροπές που εμπλέκονται στη διαδικασία της επιτροπολογίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διεθνείς πτυχές του θέματος αυτού, είναι σημαντικό να σας υπενθυμίσω ότι αν υπάρξουν και άλλες χώρες οι οποίες θα ακολουθήσουν ένα συγκρίσιμο σύστημα για την ε, εμπορία εκπομπών, θα πρέπει και εμείς να προβληματιστούμε κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συντονισμού με τις άλλες αυτές χώρες, ώστε να μπορούν και άλλες χώρες να συμμετέχουν στο σύστημά μας με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι συντονισμένος και συμπεφωνημένος και φυσικά που θα έχει αποτελέσει ε, αποτέλεσμα προηγουμένων συνεννοήσεων και εδώ πέρα φυσικά περιμένουμε να έχουμε και την άποψη των εμπειρογνωμόνων Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο φυσικά έχει διεθνείς διαστάσεις και υπήρξε και μια συνέντευξη τύπου όπου συζητήθηκε το θέμα της ε, ενσωμάτωσης των εκπομπών από, από, τις, ε, από τις πτήσεις αεροπλάνων και για το θέμα αυτό νομίζω ότι υπήρξε μια σημαντική πρόοδος, ήταν παρούσα και η κυρία Χέντεγκαρτ, υπήρξε πληροφόρηση για το θέμα αυτό. Φυσικά η κυρία Επίτροπος θα μπορούσε να μας αναφέρει και αυτά τα θέματα. Θα ήθελα όταν λάβει το λόγο η κυρία Χέντεγκαρτ να αναφερθεί και στο συγκεκριμένο αυτό ζήτημα. Θα ήταν χρήσιμο σε όλους και περιμένουμε να έχουμε και λεπτομέρειες από την Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Αυτά λοιπόν η διαδικασία όπως σας είπα είναι έχουμε χρόνο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Είναι σε δύο τμήματα η συνεδρίασή μας. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τον κύριο Σόσα Βάγνερ από την Επιτροπή Βιομηχανίας. Θα ακολουθήσει η κυρία Επίτροπος και μετά θα λάβει το λόγο εκπρόσωπος του Συμβουλίου και στη συνέχεια στο δεύτερο τμήμα θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες και θα έχουμε, πιστεύω, αρκετό χρόνο για να υπάρξει και ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Σόσα Βάγνερ. Ευχαριστώ κύριε Βάγνερ. Ευχαριστώ κύριε Γκρότερ που μου δίνετε τη δυνατότητα να λάβω το λόγο σε αυτή την ακρόαση. Είναι μια τιμή για μένα το να είμαι εισηγητής γνωμοδότησης για αυτή την έκθεση από την Επιτροπή Ενέργειας Βιομηχανίας και Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Επιτροπή την οποία εκπροσωπώ εγώ αυτό φυσικά είναι ένα θέμα ιδιαίτερο ενδιαφέροντος και είναι λογικό να είναι έτσι γιατί πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει κομικό χαρακτήρα στη βιομηχανική πολιτική και την πολιτική έναντι της κλιματικής αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξάλλου, έχει παίξει ρόλο πρωτοπόρου στην οργάνωση μιας αγοράς για τα πιστοποιητικά δικαιωμάτων εκπομπής ε, αερίων του θερμοκηπίου και άλλα τμήματα του κόσμου παρακολουθούν με προσοχή το πείραμα αυτό, την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε ποιο τρόπο μπορεί να οργανωθεί και από τη δική του πλευρά η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών. Φυσικά εγώ ως συζητητής έχω γνώση μεν του θέματος, αλλά προς το παρόν εγώ συλλέγω πληροφορίες που παίρνω από τη γραμματεία της Επιτροπής μας, τόσο της Επιτροπής ε, βιομηχανίας και ενέργειας όπως και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και επεξεργάζομαι αυτή την τεκμηρίωση που μου δίνουν οι δύο επιτροπές για να διατυπώσω την γνωμοδότηση της δικής μας Επιτροπής. Το τελικό αποτέλεσμα βέβαια της διαδικασίας στην Επιτροπή Ήτρε δεν μπορώ να το προδικάσω, θα είναι το αποτέλεσμα και της δικής μου εργασίας, αλλά και των συζητήσεων που θα λάβουν χώρα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας, τις πολιτικές ομάδες και τους σχεώδεις εισηγητές. Επομένως, από την έποψη της διαδικασίας, τα πράγματα έχουν έτσι, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. Εγώ απλώς είμαι στη φάση της ανάγνωσης και της ανάλυσης των ε, στοιχείων που μου δίνουν οι δύο επιτροπές και μετά θα περάσω τη συζήτηση με τους σκιώδεις εισηγητές και μέσω αυτών με τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Όλα αυτά μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος που μου έχει δοθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια βάσει και της δικής μας θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να οριστικοποιήσει τις θέσεις της για το ευαίσθητο αυτό θέμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να περατωθεί αυτή η διαδικασία το ταχύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα εκπομπής αριών του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά παραμένω στη διάθεσή σας για να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Αν μπορώ και να απαντήσω, αυτό θα μου δώσει μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βάγκνερ. Παρακαλώ την Επίτροπο να λάβει το λόγο και να κάνει μια εισήγηση, να μας μιλήσει όμως και για τις καινοτομίε του ΙΤΕΣ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα είναι λίγο, λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα από ό,τι με τις ε, ε, ε, ανταλλαγές εκπομπών στις αερομεταφορές. Λίγο πιο περίπλοκα. Ξέρετε, το θέμα μας απασχολήσει. Ήταν πολλέ οι χώρε, ήταν κάποιε οι χώρε οι οποίε είχαν σε έντονου τόνου ε, διατυπώσει τι αντιρρήσει του, ε, στι προτάσει μα. Ξέρετε πόσο σαφή ήταν η δική μα στάση και ξεκάθαρη. Πόσο είπαμε δηλαδή, πώς είπαμε ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση κανείς περισσότερο θα μπορούσε να επιθυμεί μια γενική ρύθμιση των περιορισμών των εκπομπών ε, από, τις, από την αεροπορία, από τις αερομεταφορές. Το θέμα αυτό οδήγησε σε ένα μακροχρόνιο δημόσιο διάλογο. Κάποιοι επεδίωξαν, κάποιες, ή περίμεναν κάποιες ενδείξεις ευελιξίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επεδίωκαν από καιρό και περίμεναν αυτά τα δείγματα ευελιξίας να δοθούν, να τους χορηγηθούν χωρίς από πλευράς τους να τροποποιήσουν κάτι τρόπο, τρόπο τη στάση τους ή τις απαιτήσει τους από την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου την προηγούμενη Παρασκευή στο Μόντρεαλ αλλά και πιο πριν συνεργαζόμαστε και προχωρούμε σε διάλογο με πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις με κράτη εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τους λέμε ότι ναι θέλουν μια παγκόσμια ε, διευθέτηση, μια συμφωνία παγκοσμίου εμβέλειας αλλά πρέπει και εσείς να βρείτε κάποιες λύσεις ώστε να μπορέσουμε από την ΙΚΑΟ να καταλήξουμε σε αποφάσεις θετικές. Και οι τελευταίες ειδήσει που έχουμε από την ΙΚΑΟ είναι ότι επιτεύχθη συμφωνία από τις μεγάλες χώρες μεταξύ άλλων, τα οκτώ ευρωπαϊκά κράτη που εκπροσωπούνται, αναπτυσσόμενες χώρες, ανεπτυγμένες χώρες του και προέκυψαν ενδιαφέροντα πράγματα από αυτή τη συνεδρία του Συμβουλίου. Καταρχάς ότι η ηγεσία της ΣΥΚΑΟ θα ε, εγκαθιδρύσει μια ομάδα πολιτική υψηλού επίπεδου ε, που θα πρέπει να ασχοληθεί με τα ζητήματα που έχουν μείνει εκρεμή, που δεν έχουν καλυφθεί, γιατί πολλά πράγματα έχουν ήδη γίνει, αναλύσεις και έχουν γίνει, και τώρα πρέπει σε επίπεδο πολιτικό υψηλού επίπεδου να προχωρήσουν τα ζητήματα. Το έχουμε ζητήσει, ήταν πολύ σημαντικό. Δεύτερο, σαφές συμπέρασμα, είναι ότι πρέπει να έχουμε τρεις πλέον βάσεις για μηχανισμούς στηριζόμενους στην αγορά με ουσιαστική ε, μία πρόταση, μέσα σε μία πρόταση που θα πρέπει να κατεθεί το στην φθινόπωρο από την ΕΚΑΟ και εν τέλει και ουσιαστικά η αλλαγή είναι ότι πλέον ρητά αναφέρεται πως και στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταγραφεί σημαντική πρόοδος για τους μηχανισμούς, Παγκόσμιο Οργανισμό Αγοράς, ε, ένα από τα κέρια αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γνωρίζετε, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εν ολίγης έγινε σημαντική πρόοδο, σημειώθηκε σημαντική πρόοδο από πλευρά τη ηγεσία τη ΙΚΑΟ, με τι πολλέ προσπάθειε που έχουν γίνει αυτό το διάστημα για πρόοδο. Και όλα αυτά είναι πολύ καλά, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο στόχο μα. Γίνονται και συνεχίζονται και θα γίνουν πολύ σκληρέ διαπραγματεύσει Γι' αυτό και σήμερα δημόσια ανεκοίνωσα ότι θα συστήσω στα κράτη-μέλη και το κοινοβούλιο σας όταν τεθεί το ζήτημα του ETS του Ευρωπαϊκού προκειμένου να αναπτυχθεί ένα θετικό κλίμα γύρω από τις διαπραγματεύσεις αυτές, εμείς να παγώσουμε το ρολόι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό ως έκφραση από τις διεθνείς ε, διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Παγώνει το ρολόι, σταματάει το ρολόι και βέβαια με κάποιο χρονικό περιορισμό, διότι θέλουμε στην προσεχή στη Γενική Συνέλευση της ΣΥΚΑΟ να φτάσουμε μέχρι και να σταματήσουμε την κουβέντα πλέον με την έννοια ότι θα έχουμε επιτύχει συμφωνία. Ουσιαστική πρόοδο στην προσεχή φθινοπορεινή σύνοδο της ΣΥΚΑΟ. Και έτσι λέμε ότι σε μια-δύο εβδομάδες θα, θα υποβάλουμε τις τεχνικές προτάσεις για το τι θα πρέπει να κάνουμε με συστάσεις προς τα κράτη-μέλη και προς το κοινοβουλίο σας. Και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκάθαρα λέμε ότι πρέπει να έχει χρονικά όρια. Αυτή η προσπάθεια μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση και αν δεν σημειωθεί μέχρι τότε πρόοδος, τότε προφανώς ξαναγυρνάμε στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Αυτομάτως. Για να συντομεύω δηλαδή και με άλλα λόγια, αυτό που λέμε είναι, κοιτάξτε τώρα σας δίνουμε μια ευκαιρία, υπάρχει μια ευκαιρία να εξασφαλίσετε αυτό που θέλετε ανέκαθεν από την Ευρώπη, δηλαδή μια παγκόσμια ε, συμφωνία για τις ε, αεροπορικές μεταφορές, αξιοποιήστε την, αλλά πρέπει και εσείς να κάνετε πλέον παιχνίδι. Και άρα θα πρέπει να εμπλακείτε στην διεθνή αυτή ε, διαδικασία η οποία ελπίζουμε πω θα στεφθεί με επιτυχία. Εμεί από πλευρά μα, από ευρωπαϊκή πλευρά, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προ το στόχο αυτόν. Σα ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να σα ενημερώσω για τι τελευταίε εξελίξει στον τομέα ε, τη ε, αεροπορία. Έχουμε βεβαίω ε, διαρκεί και σκληρέ διαπραγματεύσει με του εταίρου μα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει πλέον να στεφθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια σε επίπεδο Διεθνού Οργάνωση Πολιτικής αεροπορία, Ελπίζω θα μπορέσω να έχω την ευκαιρία σύντομα να σα ενημερώσω για νέες πρόοδους. Και τώρα θα περάσω στην ουσία της σημερινή συνεδρίασης. Σα ευχαριστώ καταρχάς για την πολύ ε, επίκαιρη αυτή ευκαιρία που δίνεται για τη μήνυα ακρόαση να συνοηθούμε και να εξηγήσουμε τι εννοούμε. έχουμε δώσει ήδη και στην Επιτροπή Βιομηχανία κάποιε ιδέε. Όταν συζητούμε τα θέματα αυτά για να ξεκινήσω, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι το ETS, το σύστημα ανταλλαγών, έχει σε τεχνικού όρου ικανοποιητικά λειτουργήσει. Μείωση των στόχων που είναι βέβαια ο κύριος, ε, η κύρια, ο κύριος σκοπός ε, δημιουργίας του συστήματος αυτού, αλλά ταυτόχρονα όπως εξήγησε και ο κύριος Πρόεδρος, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση έχει ουσιαστικά περιορίσει σημαντικά τις προτινόμενες εξαγορές ε, πιστοποιητικών πολύ περισσότερο από ό,τι περιμέναμε στην, την εποχή που θεσπίζαμε το σύστημα και ταυτόχρονα λόγω της, του αποκλεισμού των πιστοποιητικών CDM. Ξέρω ότι είχατε υποστηρίξει εσείς. δηλαδή μηχανισμού ε, καθαρής ανάπτυξης, ε, τώρα βρισκόμαστε σε μια πιο δύσκολη κατάσταση. Και έτσι η συνέπεια είναι ότι μεγάλο πλεόνασμα πιστοποιητικών εκπομπών έχει συσσωρευτεί που θα αυξηθεί εάν δεν αναλυφθεί δράση. Το πλεόνασμα αυτό δεν φαίνεται να τίνει να μειωθεί μέχρι το 2020. Και γιατί. Διότι ακόμη και αν ξεφύγουμε από την οικονομική κρίση και αρχίσει να αυξάνεται η ζήτηση για τα πιστοποιητικά, θεωρητικά με βάση την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς θα αυξηθεί και η τιμή, αλλά το πλεόνασμα θα παραμείνει στο σύστημα και άρα δεν θα δούμε αύξηση των τιμών όπως θα έπρεπε κανονικά να συμβεί. Πράγμα το οποίο θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για την, ε, τις εκπομπές ε, άνθρακα και για το μελλοντικό σχεδιασμό. Γιατί ξέρετε ότι είχαμε στόχο αρχικά να μειώσουμε τι εκπομπέ ταυτόχρονα όμω γνωρίζαμε ότι ήταν πολύ σημαντικό και να δημιουργηθούν κίνητρα για τη μετάβαση. Γι' αυτό άλλωστε και όταν συζητούσαμε την οδηγία για την αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργεια, είχαμε επικεντρωθεί στο θέμα αυτό. Άρα λοιπόν τώρα και έχει δύο φορέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωρίσει τη σημασία του θέματος αυτού με την έκθεση για, τις, για τον οδικό χάρτη για τις ε, χαμηλές εκπομπές σε άνθρακα αλλά και για την οδηγία για την αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας όπου εσείς στο Κοινοβούλιο είχατε επίμονα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει μια αναθεώρηση του λεγόμενου backloading προκειμένου να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό ETS. Και ήταν πολύ σαφής η πρότασή σας με την, ε, στην οδηγία για την αποτελεσματικότητα ενέργειας όπου λέγατε ότι θα πρέπει η πρώτη έκθεση να συνοδεύεται από μια αναθεώρηση, μια επισκόπηση της τρίτης φάσης ε, για το ETS. Αυτή είναι η δουλειά που προσπαθούμε τώρα εδώ να επιτελέσουμε και έτσι ξεκινάμε. Με μια πρόταση ε, φυλασσόμενοι ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον πίνακα, το χρονοδιάγραμμα για, τις, ε, για το backloading και με τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Προσπαθούμε λοιπόν να διευκρινίσουμε την οδηγία για το ETMS. Ο κύριος Γκλότ ε, ανέφερε ότι είναι πολύ απλή η τροπολογία, η τροποποίηση της οδηγίας συγκεκριμένα. Δεν είναι περίπλοκη, έχει πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής αυτή οδηγία μας, αυτή η τροπολογία στο κείμενο της οδηγίας και δεδομένου το κοινοβούλιο μας είχε ζητήσει να εφαρμόσουμε ή να υιοθετήσουμε καλύτερα το μέτρο του backloading, τώρα θα έλεγα ότι ελπίζουμε, στηριζόμαστε, προσδοκούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει, θα εγκρίνει αυτή την τροποποίηση ώστε να εισαχθεί αυτή η ρήτρα του backloading στην οδηγία για να μας επιτρέψει έτσι να την υλοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Βέβαια, αντιλαμβανόμεθε ότι υπάρχουν συζητήσει και σε Συμβούλιο και σε Επιτροπή για την Κλιματική και στην Επιτροπή του Κοινοβουλίου για την Κλιματική Αλλαγή, αλλά και σε επίπεδο Συμβουλίου, όπου διατυπώνονται αιτήματα και περισσότερε πληροφορίε ω προ τι συνέπειε του backloading και με προοπτική να κρατηθεί το ETS σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ελπίζω, ωστόσο, και προσδοκώ ότι η εβδομάδα αυτή με τις συστήσεις που γίνονται θα σας προσφέρει περισσότερες ε, πληροφορίες και σαφήνεια. Έτσι λοιπόν την Τετάρτη αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια έκθεση για την εξέλιξη στην αγορά άνθρακα με συνοδευτικά μέτρα. Επομένως η δεύτερη πρόταση, η δεύτερη υπόσχεση που είχαμε προβάρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο συγκεκριμένα υιοθετείται, ε, υλοποιείται με αυτή την πρόταση της ανακοίνωσης. Και επίσης συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για, τα, για τους όγκους του backloading. Ξέρετε ότι υπάρχουν τρία αριθμητικά στοιχεία που είχαν προταθεί και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιλέξει ποιο από αυτά ποια από αυτές τις ποσότητες θα προτείνει στις επιτροπές για να αποφασίσει μετά και το Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο. Στη διαδικασία αυτή την εσωτερική για λήψη αποφάσεων δεν έχουμε καταλήξει και δεν μπορώ οριστικά να επιβεβαιώσω πότε ακριβώς θα έχουμε στη διάθεσή μας για να κοινοποιήσουμε αυτά τα νέα στοιχεία. Πρέπει να πω ότι έχουμε πλησιάσει πολύ στο στόχο αυτής, της λήψης αυτής της απόφασης και ελπίζω και εσείς να αντιληφθείτε ότι πρέπει να έχουμε αυτό το χρόνο. Και βεβαίω, άπαξ και ληφθεί η απόφαση για λόγου διευκόλυνση και τη ομαλή λειτουργία τη αγορά, γιατί αυτό είναι καθήκον μα ε, για το στόχο τη ρύθμιση τη αγορά, θα ανακοινώσουμε το περιεχόμενο τη απόφαση. Άπαξ και δημοσιευθούν τα έγγραφα. Θα υπάρξει βέβαια και η υλοποίηση της ε, πρόσκλησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη των συνοδευτικών ε, μέτρων, των εκτελεστικών ε, μέτρων. Και από εκεί και πέρα θα είναι θέμα Κοινοβουλίου και Συμβουλίου να επιλύσουν το ζήτημα των ισορροπιών στήτιας. Τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Το πλεόνασμα του ενός περίπου δισεκατομμυρίου αδειών στα τέλη του 2011 σύντομα θα έχει αγγίξει τα 1,5 δις μέχρι το τέλος του 2012. Αυτό νομίζω ήδη είναι επαρκή ένδειξη ότι χρειάζεται να λάβουμε ταχύτατα δράση. Η αγορά χρειάζεται σαφήνεια, η παρατηνόμενη αβεβαιότητα δεν είναι υπεύθυνη επιλογή και χρειάζεται η αγορά απόφαση για τις ποσότητες του backloading και καταρχήν πριν από το τέλος του έτους, πριν από την έναρξη δηλαδή, της επόμενης φάσης δημοπράτησης. Και πρέπει να επιδείξουμε την πολιτική βούληση για λήψη αποφάσεων, για υλοποίηση των υπεσχημένων ταχύτατα, όπως άλλωστε είχε στήσει τον Ιούνιο το Κοινοβούλιο. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στην περιγραφή της δημοπράτησης, στην εικόνα που ήδη έχει τροποποιηθεί από την Επιτροπολογία. Θα ήθελα να σας το υπενθυμίσω αυτό ότι δηλαδή λόγω διαφόρων πτυχών που είχαν προβληθεί νωρίτερα είχαμε ήδη μια διαδικασία front-loading, προκαταβολικής δηλαδή, ε, εκχώρησης, ενώ κανείς δεν είχε αντιδράσει. Καθώς αυτή ήταν και η υπεύθυνη στάση την ε, ώρα που έγινε. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ελπίζοντα στην κατανόησή σα, ότι η πρόταση για την τροποποίηση τη οδηγία, όπω την εννοεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι μια λύση που εξετάζουμε πριν από την υιοθέτηση του κανονισμού για το backload από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλω ξεκάθαρα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την παραμικρή διάθεση και πρόθεση να καθυστερήσει, να προδικάσει ή να ε, αντιπαρέλθει το Κοινοβούλιο ω προ τη λήψη αποφάσεων στον τομέα δεν έχει την πρόθεση λοιπόν, δεν έχει μία πρόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει οριστική απόφαση για backloading χωρίς να έχει ρυθμιστεί το θέμα αυτό από εσά ως αρχή συνομοθετική. Συναρμόδια για την νομοθεσία. Και βεβαίως υπάρχουν, πρέπει να επισημάνω, ήδη ε, εγγυήσεις μέσα από την ε, διαδικασία της επιτροπολογίας ή αδίποτε τροποποίηση άπαξ και εγκριθεί από την ε, ειδική πλειοψηφία των κρατών μέλων στην Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή μέσα σε τρεις μήνες πρέπει να επικυρωθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ιδάλλως και μόνο ιδάλλως μπορεί να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τρίτη φάση. Και χρειάζεται και επαρκής χρόνος για το backloading και την αναθεώρηση του σχετικού χρονοδιαγράμματος. Θέλω δηλαδή να ξεκαθαρίσω ότι ανεξαρτήτως της διαδικασίας της συναπόφασης, τόσο το Συνοβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο έχουν και θα έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν και να παρεμποδίσουν την κρύψη αποφάσεων σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένα από την ε, προτινόμενη τροποποίηση. Μια δεύτερη πρόταση, μια δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω, ότι στις συνήθεις συνθήκες αγοράς ανταποκρίνεται η προσφορά στη ζήτηση, αλλά χωρίς παρέμβαση. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι που σας απασχολεί. Και λέτε γιατί να μην αφήσουμε την αγορά ελεύθερη να λειτουργήσει, γιατί πρέπει να παρεμβαίνουμε. Ναι, πρέπει όμω να σας πω ότι το ETS είναι όντως ένα μέσο, ένα εργαλείο στηριζόμενο συνθήκες αγοράς, αλλά λόγω των συνθήκων που επικρατούν εδώ, και θέλω να το υπογραμμίσω εδώ ενώπιον όλων σας, έχουμε να κάνουμε με ιδιαίτερες συνθήκες, με έκτακτες συνθήκες και γι' αυτό προτείνουμε λόγω αυτών των εκτάκτων συνθήκων και εξαιρετικών συνθήκων τη συγκεκριμένη ε, το συγκεκριμένο μέτρο. Δεν θα πρέπει το μέτρο να θεωρηθεί ως παρέμβαση στην αγορά, δεν θα πρέπει να παρερμηνευθεί, αφορά καταρχά ένα πολύ περιορισμένο τμήμα τη ε, οδηγίας, όχι όλες τις ε, άδειε. Εδώ μιλούμε μόνο για backloading. Σας παρακαλώ μην θεωρήσετε ότι μπορεί να επηρεάσει το σύνολο των αδειών στο σύστημα, γιατί αυτό παραμένει το ίδιο. Απλώς στα πρώτα έτη της προσεχικούς φάσεως θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να έχουμε ε, μια αντίδραση ως προς την πλημμυρίδα αδειών που αντιμετωπίζει η αγορά. Και βεβαίως, όπως είπα, τα μέτρα αυτά είναι έκτακτα. Τέταρτον και, και επόμενο θέμα, Πρόεδρε. Χρειάζεται ταχύτατα να ληφθεί απόφαση για το backloading. Είναι ένα μέτρο βράχη πρόθεσμο. Θα έχει μόνο περιορισμένες χρονικά συνέπειες και γι' αυτό πρέπει να υιοθετηθεί εγκαίρως για να μπορέσει να επαναφέρει σε ισορροπία τις αγορές. Όπως υπόθηκε και την Τετάρτη αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία απόφαση για την αγορά άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ε, εξασφαλίσει την ε, υλοποίηση ουσιαστικά αποτελεσματικών μέτρων ενώ υπάρχει ανάγκη για να δημιουργηθεί μια κάποια συνένεση αν η δράση θα καλύψει την ζήτηση, την προσφορά, αν η παρέμβαση θα είναι περιορισμένη ή όχι. Όλα αυτά θα τα βρείτε στην έκθεση για την αγορά του άνθρακα Νομίζω ότι θα έχετε όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για να διαμορφώσετε μια πλήρη εικόνα πριν από τη λήψη της απόφασής σας. Συγγνώμη, αλλά μακρηγόρησα ο λίγων, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε τι είναι το backloading και τι μάλλον δεν είναι το backloading. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου στον κύριο Κώστα Παπασταύρο. Παρακαλώ, κύριε Παπασταύρο. Hello, good afternoon to On behalf of Εξ ονόματος της Κυπριακής Προεδρίας θα ήθελα να κάνω μια κάποια μικρή παρουσίαση σχετικά με τις συζητήσεις του θέματος σε επίπεδο Συμβουλίου. Η πρόταση ε, έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον προηγούμενο Αύγουστο και μέχρι τώρα έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης από την Ομάδα Εργασίας Περιβάλλοντος ΔΙΣ στις 7 και στις 17 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών οι εθνικές αντιπροσωπείες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τις επιλογές του backloading όπως πρώτον ανησυχίε σχετικά με τη νομική βάση παρέμβασης στα πλαίσια της ρύθμιση της τιμή του άνθρακα. Δεύτερον, την πιθανή σύνδεση αυτή της αναθεώρησης με κάποια μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα δώσουν περαιτέρω εγγυήσει για τη σωστή λειτουργία της αγοράς άνθρακα. Και τρίτον, το εύρος των διακριτικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Επιτροπής μέσω της προτινόμενης τροπολόγησής τους. Στην παρούσα φάση δεν έχει καμία αντιπροσωπεία εκφράσει μια σοβαρή επιθυμία για την διεύρυνση του εύρους της αναθεώρησης έτσι ώστε να πλεράσουμε σε πλήρη μεταρρύθμιση του ETS. Σε γενικότερο επίπεδο οι εθνικές αντιπροσωπείες έχουν την τάση να συνδέουν τις συζητήσεις της προτινόμενης συγκεκριμένης αυτής ρύθμισης με τις συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν και στα πλαίσια της Επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος, για την αντιμετώπιση συνεπειών της αλλαγής κλίματος. Σημειώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαθέσιμη να αναλάβει δράση στην περίπτωση που το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ευχαριστώ και το Συμβούλιο για την παρέμβασή του. Έχουμε τώρα τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε συζήτηση. μαζί με τους σκιώδεις εισηγητέ καταρχήν και έχουμε άλλους 16 συνολικά ομιλητές. Θα πρέπει να υπάρξει συντομία στις παρεμβάσεις. Θα ήθελα όμως να δώσω καταρχήν το λόγο στους σκιώδεις εισηγητέ. Και για το ΕΛΚ η κυρία Κόρχολα, η εισηγητρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για την απόφαση την οποία πήρατε για να παγώσετε το θέμα αυτό σε σχέση με τις αερομεταφορές. Και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι μονομερείς ευρωπαϊκές δράσεις, γιατί πολλές φορές δεν βοηθούν ιδιαίτερα στα πλαίσια της αναζήτησης μιας γενικότερης λύσης στο θέμα της αντιμετώπισης των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών σχετικά με αυτό που είπατε ότι ανταποκρίνεστε στα δικά μας αιτήματα. Τι θέλουμε εμείς σαν κοινοβούλιο. Νομίζω ότι έχει υπάρξει μια υπερερμηνεία, υπερβολική ερμηνεία των προτάσεών μας. Τη στιγμή που έγιναν δεκτά τα ETS, η ιδέα του backloading δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα εξηγήθηκε επαρκώς δεν είχαμε χρόνο να αντιμετωπίσουμε τις προτάσεις οι οποίες έγιναν και παραμένουν εκκρεμότητες πριν υπάρξει εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς σαν παράδειγμα το θέμα της αλλαγής του χρονισμού των ε, πληστηριασμών συμβαδίζει με το άρθρο 9 του κανονισμού της οδηγίας μάλλον για το ETS. Λέγεται ότι ο αριθμός των δικαιωμάτων θα πρέπει να μειωθεί με γραμμικό τρόπο στην περίπτωση του backloading κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ισχύσει, οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξει θέμα με την εφαρμογή της, της ε, ε, οδηγίας. Και γενικά το Συμβούλιο δέχεται μια τέτοια πρόταση για να υπάρξει μια συμφωνία σε επίπεδο AD. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεπεράσει τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει. Και μιας και μιλάμε για το backloading, όλοι γνωρίζουν ότι ο βασικός στόχος είναι το λεγόμενο set aside. Αυτή είναι και η ερώτησή μου. Κάποια από τα επιχειρήματά σας προς αυτή την κατεύθυνση θα έλεγα πηγαίνουν. Είπατε ότι η αγορά έχει ανάγκη από διαφάνεια και έχει ανάγκη και από προβλεψιμότητα. Γνωρίζουμε ότι είναι λογικό βέβαια οι τιμές να είναι χαμηλές τώρα που η ζήτηση είναι χαμηλή. Αυτό ακριβώς είναι κάτι λοιπόν το οποίο θέτει σε αμφισβήτηση το, νομικό αίσθημα, το αίσθημα νομικής ασφάλειας θα έλεγα όταν ξαφνικά η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει ε, τα σχέδια και αυτό έχει χειροτερεύσει ε, θα έλεγα και το ευρωπαϊκό επενδυτικό κλίμα. Αυτό είναι το feedback το οποίο μας δίνουν πάρα πολλοί βιομηχανικοί τομείς, ότι με τις προτάσεις σας ε, μειώνεται την ελκυστικότητα των επενδύσεων. Βέβαια η παραγωγή ενέργειας ε, έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτήν την μηχανή παραγωγής ρευστού. Αλλά υπάρχουν άλλοι κλάδοι που ανησυχούν ιδιαίτερως για τα σχέδιά σας. Γιατί να αυξήσουμε το κόστος τη στιγμή που έχουμε ανάγκη από ανάπτυξη. Θα επανέλθω στα θέματα αυτά, πρέπει να αφήσω χρόνο και σε άλλους συναδέλφους. Chris Davis, από πλευρά των φιλελευθέρων, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για τις δηλώσεις που κάνατε για τις αερομεταφορές. Είναι καλοδεχούμενη η πρόοδος η οποία συνετελέστη, ε, γι' αυτό εσείς ο ίδιος έχετε κάνει προσπάθειες και αυτό αντικατοπτρίζει και τις συζήτησεις που κάνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο για το ρόλο μας στην παγκόσμια αγορά. Κανένα κράτος μόνο του δεν θα μπορούσε να σημειώσει την πρόοδο την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής. Μία ερώτηση. Το ε, ETS θα εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές, ε, στους ευρωπαίους αερομεταφορείς ή η κατάργηση είναι ε, σφαιρική. Τώρα για το backloading δεν είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος. Πρόκειται για ένα μέτρο θα έλεγα χωρίς συνέπεια που θα προκαλέσει σύγχυση θα πρέπει μακροπρόθεσμα εμείς να μεταρρυθμίσουμε λίγο το ETS, το ETS για να αποκαταστήσουμε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης το οποίο απαιτούν οι επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρειαζόταν να κάνει τις προτάσεις αυτές. Είχε τις αρμοδιότητες τις οποίες χρειάζεται έτσι ώστε να ρυθμίσει κάποια από τα προβλήματα αυτά χωρίς να υπάρξει ανάγκη χρήσης της διαδικασίας συν απόφασης. Γιατί δεν ακολουθήσατε αυτή την επιλογή. Μήπως δεν υπάρχει. Ευχαριστώ Chris Davis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον, την κυρία Επίτροπο για την παρουσία της και τη συμμετοχή της σε αυτή τη συζήτηση. Απλώς για τα θέματα της αεροπορίας. Είπατε ότι πρέπει να σταματήσουμε το ρολόι. Σταματήσαμε το ρολόι. Καλή, καλή έκφραση ήταν αυτή. Αλλά σταματήσαμε το ρολόι όταν η ΙΚΑΟ αποφάσισε να φτιάξει μια ομάδα υψηλού επίπεδου και πολιτικού χαρακτήρα για να μελετήσει τα θέματα αυτά. Γιατί σταματήσαμε λοιπόν το ρολόι. Και είπα θα ξαναγυρίσουμε στη δουλειά και θα αρχίσει να δουλεύει το ρολόι όταν υπάρχει πρόοδος. Αλλά πώς θα κρίνουμε το ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος. Το να σταματήσουμε τώρα το ρολόι σημαίνει ότι δεν ασκούμε πίεση στην ΙΚΑΟ, στον Οργανισμό Διεθνούς ε, Πολιτικής Αεροπορίας. Αφού λοιπόν δεν δουλεύει το ρολόι, δεν ξέρουμε τι ώρα είναι και δεν ξέρω πόσο καλή είναι αυτή η στρατηγική. Αυτά λοιπόν για την, τον αεροπορικό κλάδο. Εγώ θα ήθελα να ξέρω πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κρίνει την πρόοδο στον ΙΚΑΟ. Τώρα για το λεγόμενο backloading στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Συμφωνώ με τον Κρίς, ούτε και εγώ έχω μεγάλο ενθουσιασμό για ένα τέτοιο σύστημα, να είμαι σαφής. Και για τους συναδέλφους μου του ΕΛΚ, που στέλνουν επιστολές οι οποίες δεν ακριβώ συνάδουσες με αυτά που είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο στο παρελθόν. Και μέσα σε αυτά ήταν και το ΕΛΚ. Είχαμε ζητήσει δύο πράγματα στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Άμεση δράση πρώτον στη διαδικασία, στο προφίλ των πληστηριασμών. Άμεση δράση, αυτό σήμαινε backloading, κατεπηγόντως αν θέλετε. Και η δεύτερη αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν διαρθρωτικά μέτρα πριν φτάσουμε στην τρίτη φάση της εμπορίας εκπομπών. Αυτέ ήταν οι δύο αιτήσει που διατύπωσε το Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή εσείς μας δίνετε μία απάντηση σε ένα από τα δύο. Για το backloading. Το ότι κάποιοι αλλάζουν γνώμη στο Κοινοβούλιο δεν έχει σημασία για εσά. Αλλά τι κάνουμε με τα διαφορετικά μέτρα. Την Δετάρτη θα μας δώσετε μία έκθεση σε σχέση με την αγορά διοξιδίου του άνθρακος, άνθρακος ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε πώς θα είναι Δύο δισεκατομμύρια πιστοποιητικά χωρίς αν δεν υπάρξει κάποια δράση. Το backloading από μόνο του δεν θα αλλάξει τίποτα. Είναι απίθανο να δράσει η αγορά και να αντιδράσει εάν δεν κάνουμε τίποτα να αντιμετωπίσουμε αυτό το διαφθορτικό πλεόνασμα για τις άδειε εκπομπών. Ίσως την Τετάρτη θα δώσετε κάποιες προτάσεις για έξι δυνητικά μέτρα. Τι θα γίνει μετά όμω, πάλι φάση διαβούλευση για όλα τα κράτη-μέλη που ξέρουμε ποια είναι η θέση του. Η Πολωνία δεν θέλει να κάνει τίποτα. Η... Το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να πάει στο μείον 30. Θέλουμε άλλο ένα γύρο λοιπόν διαβούλευση. Κάνατε ανακοινώσει, οδικού χάρτη, επισκοπή. Όλοι ξέρουν ποιε θέσει έχει ο καθένα. Χρειαζόμαστε μια πρόταση από την Κομισιόν ώστε να παγιώσουν οι χώρε, όλε οι χώρε, τη θέση του. Ξέρουμε για την Πολωνία και την Αγγλία. Δεν ξέρουμε για τη Γερμανία όμω. Τι θα πει η Γερμανία δεν προτείνει κάτι συγκεκριμένο η Κομισιόν, τότε τελικά θα καθορίσει τη θέση της. Δεν βοηθάει μια περαιτέρω διαδικασία διαβούλευσης. Τι θα κάνει αυτή η διαδικασία διαβούλευσης για τις έξι προτάσεις σας που θα δώσετε την Τετάρτη στη δημοσιότητα. Όλοι ξέρουμε τι θα κάνουν. Θέλω το χρονοδιάγραμμά σας ως Κομισιόν. Πότε θα προτείνετε τα διαφορετικά μέτρα τα οποία είναι δική σας προτίμηση και να περάσετε σε πραγματική δράση. Δεν θέλω άλλη φάση διαβούλευση. Φτάνει πια. Ευχαριστώ Μπάς. Και εγώ ήμουν έτοιμο να παγώσω το χρόνο για να μπορέσετε να τελειώσετε το χρόνο σας, αλλά παρακαλώ αυτοσυγκράτηση στο, στους άλλους ομιλητές. Ο, ο, ο κ. και έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είμαι σκιώδης συγητής από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και από την Επιτροπή Βιομηχανίας αυτό τον, ε, αυτήν την ιδιότητα παίρνω το λόγο. Η κυρία Επίτροπος μας διαβεβαίωσε ότι όλα θα πάνε καλά. Πρέπει όμως να πούμε πως οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημαίνουν ότι δεν υλοποιούνται αυτά που είχαμε προβλέψει το 2008. και ότι μας ζητάτε να ε, παθεθεί το σύστημα ε, από εδώ και μπρος στα χέρια κάποιων πολιτικών να το καθοδηγήσουν με συνέπεια αποφάσεις τεχνικού χαρακτήρα, διαχειριστικές αποφάσεις, να επιφέρουν επιπλέον κόστος σε ύψος δισεκατομμυρίων ευρώ με πολύ αμφίβολα αποτελέσματα. Για δε την πρόταση για πάγωμα των ε, ποσοτήτων αυτών 400, 800 και ένα δισεκατομμύριο, 400 εκατομμύριο και 1,2. Ε, τι είδου ε, συνέπειες μπορούμε να περιμένουμε. Και ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο αφορά περισσότερο τη γραμματεία της Επιτροπής. Έχουμε ένα πλαίσιο όπου λέγεται για ορισμένου συγκεκριμένους βιομηχανικού κλάδους Αναφέρεται καταρχήν η κατάσταση των ιδρυμάτων ή των καταπιστευμάτων που χαρακτηρίζονται ως αμφισβητείες της κλιματικής αλλαγής ή αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Εδώ αναφέρεται στο κείμενο αυτό ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει εξ των αυτών που υποστηρίζουν την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ τον κύριο Σιμάνσκι. Ο κύριο Χίμπνερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καταρχήν, είπατε ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών το οποίο λειτουργεί πολύ καλά. Γιατί να το αλλάξουμε τότε. Η πρότασή σας βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να εφαρμόσει το χρονοδιάγραμμα που θέλει κατά το ΔΟΚΟΥΝ να κάνει λοιπόν το, front, το backloading έναντι, ενάντια στις ε, λειτουργίες της αγοράς, αυτό αντιτίθεται στην πραγματική εμπορική λειτουργία του συστήματος και αυτό μειώνει και υποσκάπτει την αξιοπιστία του στα μάτια των επενδυτών γιατί να δώσουμε στην Κομισιόν μια επιταγή ελευκό για να κάνει ό,τι θέλει σε σχέση με το σύστημα αυτό εν ώψη των συνθήκων που παρουσιάζονται. Κατά την άποψή μου, η Κομισιόν θα πρέπει να έχει μια δυνατότητα να παρεμβαίνει στην αγορά. Λέτε ότι πράγματι ορισμένε φορές μπορεί οι τιμές να είναι πάρα πολύ ψηλέ για τα πιστοποιητικά. Αλλά αυτό δεν φαίνεται ότι θα προκύψει με τις ε, βραχυχρόνιες αλλαγές που θέλετε να εφαρμόσετε στους πληστηριασμούς. Γιατί σας λέω ότι με τον τρόπο αυτό θα χάσουν οι επενδυτές κάθε εμπιστοσύνη στο σύστημα αυτό. Δεν νομίζω ότι μέχρι τώρα υπήρχε κάποια ιδέα για να αλλάζει το χρονοδιάγραμμα των πληστηριασμών εκπομπών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή προσεγγίζει το στόχο του 20%, έχει το στόχο του της μείωσης 20% για το 2020. Αλλά όταν ένα παιδί έχει κολλήσει γρήπη, δεν του δίνουμε αμέσω αντιβιωτικά. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι στην αγορά. Ο κύριος Σιμάνσκι. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η άποψή μου είναι παρόμοια με τους προλαλήσαντες. Νομίζω το να προσπαθήσει κανείς ε, το σύστημα αυτό με τον τρόπο με τον οποίο προτείνεται δεν είναι πολύ σωστό γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα το οποίο γίνεται αντικείμενο θα έλεγα μέχρι τώρα μια σωστής διαχείρισης και δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς ποιες είναι αυτές οι έκτακτες συνθήκες τις οποίες αναφέρεται ο κύριος, αναφέρθηκε και ο κύριος Σιμάνσκι. Πρόκειται για κάτι το οποίο θα αποσταθεροποιήσει το σύστημα, θα δημιουργήσει ε, βλάβη θα έλεγα στις ε, περιβάλλουσες οικονομικές και επενδυτικές συνθήκες. Εμείς ε, στη χώρα μου έχουμε μια πολιτική στον τομέα αυτό της εκπομπής καυσαερίων που ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες. Ε, στις προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει νομίζω ότι θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Δεν είναι σαφές λοιπόν τι θα γίνει και με το θέμα της χρηματοδότησης των περιβαλλοντικών μέτρων μέσω των προτάσεων αυτών οι οποίες ε, έχουν σαν στόχο να αλλάξουν την πολιτική η οποία υπάρχει στην Ευρώπη. Η κατάσταση λοιπόν των προτάσεων δεν είναι σαφής και αυτά τα μέτρα όχι μόνο θα δημιουργήσουν προβλήματα στην ίδια την αγορά αυτή αλλά και στην γενικότερη οικονομική δραστηριότητα. Ε, ε, Κυρία Επίτροπε, Καταρχάς ω προς την ε, διαδικασία. Προσπαθείτε να μας καθησυχάσετε παρουσιάζοντας τα πράγματα πιο ε, ήπια. Αλλά θα ήθελα να πω ότι εκφράζεται ουσιαστικά μια βούληση να ε, μπουν στο περιθώριο το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσει όπω τι επιθυμείτε. Σήμερα προσπαθείτε να μα παρουσιάσετε την κατάσταση κάπω διαφορετικά, αλλά θεωρώ ότι επιδιώκεται να εξασφαλίσετε μια σχεδόν μόνιμη μορφή εξουσία Χωρί πλαισίωση για τον προσδιορισμό των τιμών. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να φαίνεται αυτό άξιο εκπλήξεως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε μιλά για ελευθερία τη αγορά, για ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, απρόσκοπτη λειτουργία τη αγορά και βλέπω να τίνει προ την ελευθερία κατεύθυνση τώρα. Με καταπλήσετε. Ε, Ω προ την ουσία, θα ήθελα να πω ότι με τρομάζει κάπω η αβεβαιότητα δικαίου η οποία προξενείται από την επιλογή σα διότι κανείς δεν θα γνωρίζει ουσιαστικά το τι προκύπτει ως προς τις τιμές της ενέργειας σε μια χρονική στιγμή όπου και σε περίοδο κρίσης προφανώς δεν είναι ευκταίο να αυξηθούν οι τιμές της ενέργειας. Και μάλιστα ενώ μειώνονται οι τιμές της ενέργειας στις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, η πρόταση για απόφαση η σχετική με το backloading μας φαίνεται ως μια περιττή απόφαση, ένα μέτρο υπερβολικό που μπορεί και να παρακολύσει τις εξελίξεις και τις επενδύσεις πάνω απ' όλα στην Ευρώπη. Μου φαίνεται μάλιστα επιβλαβές στο χρονικό αυτό διάστημα και εις βάρος της βιομηχανίας να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τιμές γιατί προτείνεται βεβαίως μια κατώτατη τιμή, αλλά όχι και μέγιστο όριο μέσα σε μια συγκεκριμένη ποσόστοση. Ένα τέτοιο μέτρο λοιπόν χωρίς ανώτατη το επίπεδο για τις τιμές του άνθρακα θα οδηγούσε σε, μια, σε έναν εκτροχιασμό του συστήματος με πολύ σημαντικό κόστος στην ποσόστοση και επιβλαβείς συνέπειες για τη βιομηχανία μας η οποία ξέρουμε πόσο πολύ δοκιμάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τρέχουσα εποχή. Άρα δεν νομίζω ότι μπορείτε να μας πείτε πως η αύξηση στην τιμή του άνθρακα μπορεί να είναι η καλή λύση αυτή την εποχή. Ενώ, και τελειώνω πρόεδρε, θα πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα και να μην αποδυναμωθούν, τουλάχιστον οι επιχειρήσεις με πολύ υψηλέ τιμές για τον άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ για τα δύο λεπτά, λέει ο Πρόεδρος. Κύριος Κλάμερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Μια διαδικαστική ερώτηση. Από αυτά που είπε η κυρία Χίλντεγκάρτ, δεν κατάλαβα ξεκάθαρα πότε ακριβώς θα κληθούμε να δούμε μια τελική πρόταση για απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σέβεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την, ε, το δικαίωμα για συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ναι ή ου. Θα γίνει η επιτροπολογία πριν το Κοινοβούλιο να καταλήξει με την τοποθέτησή του, ναι ή ου. Γιατί δεν ήταν σαφής η ου γιατι δεν ηταν σαφη η κατασταση Και ω ε, ερετό εκπρόσωπο των πολιτών δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν σε ένα θέμα τόσο σημαντικό όπως η περιβαλλοντική πολιτική να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να τηρούνται αυστηρά οι διαδικασίες. Και γι' αυτό θα ήθελα όταν πρόκειται να γίνουν οι εσδήποτε αλλαγέ σε ένα τόσο κεντρική σημασία σου αυτό που σχετίζεται με την προστασία του κλίματος, δεν είναι δυνατόν να παραγωνίσετε το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, πρέπει να πω ότι με κατέπληξε η ανακοίνωση αυτή που εκδόθηκε σήμερα το μεσημέρι για την ε, καθυστέρηση στο θέμα της ε, πολιτικής αεροπορίας, την οποία παρουσιάζεται ως επιτυχία. Ουσιαστικά πρόκειται για επιτυχία για τα άλλα κράτη. Η Ινδία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, αυτοί κερδίζουν τον αγώνα, αυτοί που πιάζαν τόσα χρόνια. Και Είμαι διατεθειμένος να στοιχηματίσω οτιδήποτε, ότι δεν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε την παραμικρή πρόοδο σε επίπεδο ΙΚΑΟ μέχρι του χρόνου, μέχρι το προσεχές φθινόπωρο. Πολύ ευχαριστώ. Όποιο στοίχημα θέλετε, είμαι διατεθειμένος να δώσουμε ένα ραντεβού και να ξαναδούμε τι εξελίξεις θα έχουν σημειωθεί μέχρι τότε. Για να επανέλθω όμω στο backloading, το κόστο για τη μείωση των εκπομπών για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, γιατί η σημερινή ανακοίνωση για τι αεροπορικέ εταιρείε αναφέρεται αποκλειστικά σε ε, πτήσει εντό και ε, από και προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή πάλι έχουμε αυτό το επιπλέον κόστο για τι ευρωπαϊκέ ε, πτήσει. Το ίδιο και με το γενικότερο σύστημα ETS. Γιατί συνεχίσουμε να συζητούμε τέτοιες λύσεις για την προστασία της κλιματικής αλλαγές, όταν δεν γνωρίζουμε τι θα προκύψει από την Τόχα. Δεν πρέπει πλέον να αναγνωρίσουμε ότι δεν πρόκειται να μετατραπεί σε μια ε, παγκόσμια αγορά των ε, πιστοποιητικών άνθρακα ή η, η παγκοσμια οικονομία, και πρέπει να βρούμε διαφορετικές λύσεις. Ευχαριστώ κύριο Ζήμπερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο. Η απόφαση που μας παρουσιάσετε για την πολιτική αεροπαρία είναι μάλλον ένα κακό δείγμα και μια κακή, ένα κακό μήνυμα. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα πρέπει οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί να τηρούνται κιόλα. Για τα όσα είπε ο Σέφρος Μπακάιτο για την επιστολή και γιατί και εγώ την προσυπογράφω Θέλουμε πάνω απ' όλα να διαφυλάξουμε την ακαιρεότητα τη δημοκρατική διαδικασία, όπω ξεκάθαρα είπε ο κύριο Κράμερ, γιατί δεν είναι σαφέ το τι είδου αποφάσει και πώ θα ληφθούν οι αποφάσει αυτέ. Πρώτα με το ETS, μετά με το backloading. Δεν βλέπουμε δηλαδή να πρόκειται για μια μικροτροπολογία στο σύστημα του ETS, αλλά για μια ουσιώδεστατη αλλαγή στο σύστημα του ETS. Και εδώ πρέπει το Κοινοβούλιο να συμπράξει πλήρω, να συμμετάσχει πλήρω. Επίση, και χωρίς να θέλω να επιβαρύνω συναισθηματικά το όλο σύστημα, εάν κοιτάξουμε το σύστημα ETS, ε διαπιστώνουμε ότι έχει ακολουθήσει το σχεδιασμό του στη λειτουργία του αυτό το ETS. Ε Έχουμε δηλαδή βρει λύσεις οι οποίες είναι οικονομικά πιο ε, ανεκτές και τώρα αν πούμε ότι πρέπει να τα αλλάξουμε όλα αυτά και να πούμε δεν αρκούν, είναι σαν να λέμε ότι το φάρμακο δεν είναι αρκετά πικρό και πρέπει να το πικρύνουμε περισσότερο, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τι ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν θα πρέπει βεβαίως να στείλουμε εσφαλμένα μηνύματα στο βιομηχανικό κλάδο διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να διαφυλαχθεί αδίποτε επένδυση γίνεται με επίκεντρο την Ευρώπη. Γιατί λοιπόν μια επιχείρηση να φύγει έχοντας ε, ανησυχία λόγω του ETS ενώ μπορεί να έχει στη διάθεσή της με, ε, με χαμηλά με χαμηλές τιμές για τον άνθρακα, στη διάθεσή της το ποσό αυτό το αντίστοιχο ως να το χρησιμοποιήσει σε επενδύσεις μέσα στην Ευρώπη. Και τελικά το ερώτημα είναι τι επιδιώκετε. Θέλετε να είσαστε η υπερ, η υπέρ, η σούπρα αριθμιστική αρχή για το ETS ή θέλουμε να διαφυλάξουμε το παλιό σύστημα με το, με το 20% το οποίο λειτουργεί. Αν θέλουμε όμως να ανταλλάξουμε το σύστημα αυτό από την άλλη, θα πρέπει το, το κοινοβούλιο να διδραματίσει έναν ουσιώδη ρόλο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που τηρήσατε τα δυο σας λεπτά. Η κυρία Μαγιόρταν, παρακαλώ. Δύο λεπτά επίσης, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο. Και εγώ ανησυχώ όπως και άλλοι συνάδελφοι. Ανησυχώ λόγω της διαδικασίας συναπόφασης, του σεβασμού της διαδικασίας αυτής. Θέλουμε να υπάρξει αυτή η δημοκρατική διαδικασία της συναπόφασης και δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε τη δημοκρατική διαδικασία στην ανάγκη κατεπίγουσας δράσης. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η νομοθετική, σωστή νομοθετική διαδικασία για το backloading και μετά να έρθουμε στις άλλες προτάσεις της Κομισιόν. Βάσει της νομοθεσίας που είναι ήδη ενισχύει, θα πρέπει να τηρηθεί και η οδηγία που έχει να κάνει με την ενεργειακή απόδοση. Αυτή η οδηγία μας υποχρεώνει να συζητήσουμε για τα θέματα των πιστοποιητικών εκπομπών, όχι απλώς να τα αφήσουμε κατά μέρος. Εσείς λέτε συνέχεια ότι δεν έχουμε επιτύχει, δεν έχουμε βελτιώσει την κατάσταση σε σχέση με τους στόχους μας. Δεν είμαστε κοντύτερα στο να τους επιτύχουμε. Αν ακολουθούσαμε τη δική σας γραμμή, θα γινόταν πιο πολυδάπανη η ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο θα σήμαινε ότι και ο καταναλωτής θα έπρεπε να καταβάλει μεγαλύτερο τίμημα για την ενέργειά του, συγκεκριμένα τα νοικοκυριά. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά <clears throat> την αεροπορία. Συμφωνώ μαζί σας, είναι κρίμα που η Ευρώπη δεν ακολούθησε την ε, γραμμή αυτή που έπρεπε να ακολουθήσει λόγω ορισμένων υποσχέσεων που είχαν δοθεί. Εγώ νομίζω ότι στον τομέα των, ε, του αεροπορικού κλάδου δεν ακολουθήσαμε μία γραμμή που ακολουθήθηκε στο υπόλοιπο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επίτροπο για την παρουσίασή της. Θέλετε να κλείσετε, να σταματήσετε το ρολόι, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί η αγορά. Το backloading θα φέρει μονάχα μια βραχυχρόνια ανακούφιση. Αυτό είναι κάτι που είναι σαφές και έχει φανεί και από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Τελικά το αποτέλεσμα θα είναι μόνο πρόθεσμα και παροδικά να δώσει μια ανακούφιση, αλλά δεν αποτελεί αυτή η λύση καμία διαφορετική λύση. Ποιο είναι λοιπόν το χρονοδιάγραμμα για να τροποποιήσετε τον παράγοντα γραμμικής μείωσης, γιατί αυτή θα πρέπει να είναι η πρόταση της Κομισιόν. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που αναφέρθηκε από ένα από τους συναδέλφους είναι ότι το σύστημα πρέπει να διατηρήσει την αξιοπιστία του. Αν συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε συνέχεια θα θεωρούν όλοι ότι το σύστημα αυτό θα υπόκειται σε συνεχείς παρεμβάσεις από την Κομισιόν και θα χάσει την αξιοπιστία του. Επανέρχομαι στα θέματα των, της αεροπορίας. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό το μορατόριο που έχει συμφωνηθεί, ποιες πτήσεις καλύπτει και ποια αεροδρόμια προέλευσης και προορισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κυλακάκης τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το CDM, Clean Development Mechanism. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, γιατί είχαμε ζητήσει όταν είχε ξεκινήσει αυτή η υπόθεση, το σκάνδαλο αυτό το CDM, να σταματήσει να λειτουργεί. Δεν σταμάτησε αμέσως να λειτουργεί και τώρα βλέπουμε ότι έχει συνέπειες και οι συνέπειες αυτές είναι ότι πληρώνουμε πολύ φθηνά υπερβολικά φθηνά πιστώσεις, αυτό που ζητάτε τώρα με το overload, και επίσης λέγεται ότι προσπαθούμε να έχουμε και μια βιομηχανική πολιτική. Εάν θέλουμε να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική για το περιβάλλον, για τα ανανεώσιμα, για τις ανανεώσιμες πίσεις κτλ, εξυπηρετούμε ουσιαστικά την Κίνα, η οποία αυτή τη στιγμή, από ό,τι μας λένε και οι παραγωγοί, των φωτοβολταϊκών πλακών επιδοτεί προκειμένου να χτυπήσει την αγορά των φωτοβολταϊκών. Και αυτό που θα έλεγα είναι ότι βρισκόμαστε σε πολύ πολύ δεινή θέση ω προ την κλιματική αλλαγή. Να σα εξηγήσω λοιπόν με τα μέτρα σα τι συνέπειε θα έχουμε στην Ελλάδα. Θα αυξηθούν οι τιμέ ηλεκτρική ενέργεια. Ο κόσμο δεν θα μπορεί να καταβάλει το τίμημα. Δεν θα μπορεί η εταιρεία ηλεκτρισμού να επενδύσει σε νέα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Θα συνεχίσουμε με τις παλές εγκαταστάσεις να εκπέμπουμε ρήπους στην ατμόσφαιρα, πληρώνοντας ταυτόχρονα ακριβά, εμείς και οι πολίτες μας, τις πιστώσεις. Αυτό θέλετε πραγματικά να κάνετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μαγκέιβαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω αρχίσει να ανησυχώ γιατί πολλοί λένε δεν θέλουν να γίνει αυτό, δεν θέλουν να γίνει το άλλο, αλλά το θέμα είναι τι θέλετε να γίνει. Υποστηρίζετε το ETS, ξέρουμε το τι λέγατε κυρία Κόρχολα από το 2008. Οι πιο πολλοί όχι, βέβαια κάποιοι από εσά τα υποστηρίζουν. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με το ETS. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία προσπαθεί να λύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία εμείς έχουμε δημιουργήσει σαν νομοθέτες μέσω των επιμέρους παρεμβάσεων και αλλαγών τις οποίες έχουμε κάνει. Πρέπει λοιπόν συνάδελφοι να μας πείτε τι θέλετε εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλετε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά για τους συναδέλφους. Κάποιοι συνάδελφοι λένε επίσης ότι δεν είναι οι προτάσεις σας αρκετές και η δική μου κυβέρνηση το λέγει αυτό άλλωστε. Κάποιες χώρες μέλη ε, θέλουν να ξεπεράσουν τον μέσο όρο θα έλεγα τον οποίο προτείνει το Συμβούλιο. Υπάρχει ελπίδα πραγματικά να λειτουργήσει και να έχουμε κέρδη από το ETS γιατί πολλοί λένε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο και δεν σας στηρίζουμε. Κάποιοι πιστεύουν ότι δεν θα στηρίξουμε τις προτάσεις σας, οπότε και αυτοί δεν σας στηρίζουν γενικότερα και δεν ξέρω τι θα μείνει από όλη αυτή την ιστορία αν αυτές οι δύο αντιλήψεις ε, οι οποίες κρατούν σήμερα θα βοηθήσουν το ETS, θα λειτουργήσει το ECS και τι συνέπειες θα έχουμε σε επίπεδο κλιματολογικής πολιτικής. Αν δεν έχουμε μια λειτουργική αγορά στον τομέα του άνθρακα πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Ακούσαμε και για τις αερομεταφορές. Κατανοώ την Επίτροπο, πιέζεται πάρα πολύ Ελπίζω να διορθωθεί η κατάσταση και δεν είμαι πολύ αισιόδοξη γιατί γνωρίζω ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν πολλοί που θέλουν να μειώσουν την ευρύτητα της πολιτικής μας. Τώρα με τη δεύτερη εντολή Ομπάμα στις Ηνωμένε Πολιτείε γεννιούνται καινούριε ελπίδες ενώ εμείς με αυτά που λέμε σήμερα κάνουμε το αντίθετο. Ευχαριστώ κυρία Μαγκαβέν. Ο Ρέστερος έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Επίτροπος ή ζει στον Άρη ή δεν ξέρει τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προτάσεις της όχι μόνο δεν διευκρινίζει την οδηγία ETS, αλλά την τροποποιεί με τέτοιο τρόπο και παίρνει τις αρμοδιότητες να παρεμβαίνει ρυθμιστικά στην ελεύθερη αγορά, ζητώντας μια λευκή επιταγή ουσιαστικά για οποιοδήποτε μέτρο, ακόμα και με αναδρομική ισχύ. Αν περάσουν οι προτάσεις αυτές, το ETS δεν θα είναι πλέον ένα μέσο της αγοράς, θα είναι ουσιαστικά ένας ευρωπαϊκός φόρος για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Με τις τιμές αυτή τη στιγμή της ε, της συγκεκριμένης δραστηριότητας πάρα πολύ χαμηλές λόγω των μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι που θα αυξήσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, θα τις οδηγήσει σε τρίτες χώρες όπου δεν υπάρχουν κανόνες ή δεν επιβάλλονται οι κανόνες. Είμαι κατά λοιπόν της αντίληψης που έχει για την αγορά ETS Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάτι που μας βγάζει πέραν από τη λογική της δημιουργίας του και μοιάζει με τα πενταετή οικονομικά προγράμματα των Κινέζων και των Σοβιετικών. Εδώ θα συμφωνήσω με τη Μακάβαν λέγοντας ότι η πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος ασκείται ε, σφαιρικά, συνολικά, όχι μονομερός στην Ευρώπη, αποκλείοντας ή οδηγώντας μάλλον στις τρίτες χώρες τις επιχειρήσεις μας. Ο Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα θέματα των, ε, της αεροπορίας. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει κάποια νομοθεσία για τα θέματα αυτά. εγώ μπορώ να θεωρήσω ότι αυτά που έχουν γίνει μέχρι την, με τον ΙΚΑΟ, τον Διεθνέ Οργανισμό Πολιτική Αεροπορία, να τα κρίνουμε θετικά, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να αποφύγουμε τι ε, στρεβλώσει του ανταγωνισμού. Γιατί εμεί όμω κάνουμε μια, ε, ένα μορατόριο για ένα χρόνο, όταν ουσιαστικά το πρόβλημα αφορά μονάχα έξι μήνες. Ίσως θα μπορούσε να ήταν μικρότερη η αναβολή. Για το backloading, Υπάρχουν φυσικά διαφορετικές απόψεις στις πολιτικές ομάδες για το θέμα αυτό. Εγώ βλέπω θετικά αυτή την πρόταση και περιμένω και την συγκεκριμένη πρόταση από την κυρία Επίτροπο για να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποια είναι τα σχέδια της Κομισιόν, ποια είναι η έκθεση αντικτύπου στην αγορά άνθρακος και με τα στοιχεία αυτά μπορούμε να κρίνουμε ποιε θα είναι οι συνέπειε όταν έχουμε όλε αυτέ τι διευκρινήσει από τη δική σα πλευρά. Και μπορώ να σα πω ότι μέχρι στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει τις προτάσεις της Κομισιόν. Έχουμε συμφωνήσει για μια διαδικασία σε δύο στάδια για την ενεργειακή απόδοση. Καταρχήν λοιπόν θεωρούμε ότι η κατεύθυνση που ακολουθείται είναι η σωστή. Και είναι ακριβώς αυτή η γραμμή που συμφώνησε το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή για την Ενεργειακή Απόδοση. Κυρία Βάσκη Έρμπερ μου ζήτησε να θέσω ένα ερώτημα εξ ονόματος της επειδή δεν θα μπορούσε να έρθει εδώ. Αυτή υποστηρίζει μέσα σε στενά όρια το backloading αλλά πρέπει, λέει, να λάβουμε υπόψη και το λεγόμενο carbon leakage, δηλαδή τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων. Και εξάλλου Όλα αυτά που συζητάμε τώρα δεν τα συζητάμε σε κενό αέρος. Θέλουμε να υπάρξουν οι απαραίτητες ε, ρυθμίσει, αλλιώ τα κράτη-μέλη θα πάρουν μεμονωμένα εθνικέ αποφάσει. Και αυτό είναι το χειρότερο για την εσωτερική αγορά που μπορεί να προκύψει. Ευχαριστώ. Έχουμε φτάσει στο τέλο του πρώτου γύρου ερωτήσεων, λέει ο κύριο ε, Κρότερ. Για την αεροπορία ήταν πάντα πρόθεσή μας να υπάρξει μια ρύθμιση. Και από την πλευρά αυτή η Επιτροπή μας χαιρετίζει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια μηνύματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια διεθνή υποστήριξη και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει μεγάλη σημασία για το Κοινοβούλιο. Μπορεί κανείς να θέσει ό,τι είδου συστήματα θέλει, αλλά θα πρέπει να δούμε από την άλλη πλευρά τι κάνουν οι διεθνείς μας εταίροι και να τους δώσουμε ένα μήνυμα ότι από τη δική μας πλευρά μέσω της νομοθεσίας μας θέλουμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση που αναφέρθηκε σήμερα. Όλα αυτά που κάνουμε θα πρέπει να συνάδουν με τις αποφάσεις να ληφθεί υπόψη και η αεροπορία στα θέματα της, ε, το, της εμπορίας εκπομπών και από την πλευρά της, ε, τη δική μου, εγώ είμαι ο εισηγητής για τα θέματα αυτά του backloading. Και εγώ ακολουθώ απόλυτα αυτά τα οποία έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει ζητήσει κατ' επανάληψη το Κοινοβούλιο να υποβάλει η, πρόταση, η Κομισιόν μια φιλόδοξη πρόταση για τα θέματα αυτά. Και τελικά το θέμα της ε, κλιματικής αλλαγής δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί χωρίς μια εταιρική ε, αντιμετώπιση από όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά όπως είπε ο Πέτερ Λίζε, αν κατακαιρματίσουμε την πολιτική μας σε 27 εθνικές πολιτικές, τότε θα κοστίσει πάρα πολλά χρήματα αυτό και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε. Γι' αυτό αν θέλουμε να υπάρξει μια μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος, θα πρέπει να επιζητήσουμε μια προσπάθεια όσο δυνατόν περισσότερο σε διεθνές επίπεδο. Πιστεύω ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου έχει ακολουθήσει ακριβώς αυτή τη γραμμή να προχωρήσουμε με μια σταδιακή και βαθμία διαδικασία. Αυτό λοιπόν προτείνουμε και νομίζω ότι αυτά που είπε σήμερα ενώπιό μα η κυρία Επίτροπος ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο. Αλλά φυσικά σας, σε εσάς απευθύνθηκα λοιπόν και θέλω να σας δώσω το λόγο για τον πρώτο γύρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς για τις αερομεταφορές. Βρισκόμαστε στην φάση που θα έπρεπε να είμαστε σε επίπεδο των διεθνών ρυθμίσεων για τις εκπομπές. Όχι βέβαια. Αλλά είμαστε μήπως σε ένα σημείο που για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια υπάρχει πράγματι η δυνατότητα να υπάρξει πρόοδο σε διεθνές επίπεδο. Εδώ η απάντηση είναι θετική και αυτό είναι κάτι συνδέεται με αυτό το οποίο είδαμε να γίνεται στις 9 Νοεμβρίου, την προηγούμενη Παρασκευή. Αυτό δεν έπεσε από τον ουρανό. Οι δυνατότητες αυτές μας δίδονται γιατί κάποιοι δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά έτσι ώστε η δυνατότητα αυτή να γίνει πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να διακινδυνεύσουμε, να υπονομεύσουμε αυτήν την εξαιρετική ευκαιρία που έχουμε μετά από πολλά χρόνια για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για την διεθνή ρύθμιση των εκπομπών του Σάρα Μεταφορές. Θέλετε εμείς να, να δώσουμε εμείς πάσα στους αντιπάλους μας θα, έφελα, θα έλεγα μέσω ακριβώς αυτών των περιφερειακών ρυθμίσεων κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις διαπραγματεύσεις και θα χαράσει το κλίμα. Νομίζω ότι καλό θα ήταν λοιπόν να πούμε ότι δεν σας άρεσε το πρώτη, προτινόμενη ρύθμιση, αλλά παρόλα αυτά ισχύει η ρύθμιση αυτή και υπάρχει η δυνατότητα να πετύχουμε αυτό το οποίο είχαμε. Γιατί όταν είπαν ότι διαφωνούσαν, είπαν ταυτόχρονα ότι ήταν υπέρ της διεθνούς ρύθμισης και αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι να τους πάρουμε τις μετρητής και να πούμε ότι πράγματι η δυνατότητα αυτή ισχύει, είναι ανοιχτή. Και κατανοώ και ποια είναι και η θέση του ΙΚΑΟ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ξεκάθαροι ότι εμένουμε σε αυτή την θέση, αλλά ρυθμίζω κιόλα και το είπα ήδη ότι αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, αν οι χώρες αυτές, οι υπόλοιπες χώρες δεν θα έλεγα φτάσουν στο σημείο το οποίο θα θέλαμε εμείς, αυτό που είδαμε να γίνεται την προηγούμενη Παρασκευή στο ΙΚΑΟ, τότε αυτόματα, χωρίς καμία περισσότερη συζήτηση, θα επανέλθουμε σε αυτό το οποίο ισχύει σήμερα. Θα επιβάλλουμε δηλαδή την ισχύουσα ρύθμιση. Κατανοώ ότι αυτά είναι, θα έλεγα, καινούργια στοιχεία, λίγες ώρες τα έχουμε στη διάθεσή μας, το καταλαβαίνω αυτό, αυτό δημιουργεί θέματα. Αλλά παρόλα αυτά παρακαλώ να εξετάσετε τις προτάσεις αυτές, είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να υπάρξει μια διεθνή συμφωνία σε ένα τομέα όπου η Ευρώπη ήθελε να προωθήσει την πολιτική αυτή και στην ουσία παραιτηθήκαμε περιμένοντας το ΙΚΑΟ. Το ΙΚΑΟ τώρα προχωρά. Είναι μια αφορμή και ευκαιρία για μας. Για την κυρία Κόρχολα και για τον πρόεδρο. Δεν έχω βέβαια πάρα πολύ χρόνο και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες απαντώντας σε όλους προσωπικά. Αλλά για την κυρία Κόρχολα. Είπε η κυρία Κόρχολα ότι το backloading και το set aside είναι το ίδιο πράγμα και άλλες τέτοιες προτάσεις μοιάζουν με αυτά τα δύο. Όχι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο, το backloading, εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με την τροπολογία την οποία έχετε μπροστά σας. Για το set aside, το μόνιμο set aside, προφανώς θα υπάρξει συναπόφαση και τίποτα δεν θα αλλάξει αν δεν υπάρξει άποψη και από πλευράς ε, του Κοινοβουλίου. Η κυρία Κόρχολα είπε γιατί να συζητάμε το backloading όταν ο στόχος είναι το set aside. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο εμείς προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο και αυτό ε, είναι απάντηση και για το buzz στην ουσία είναι ότι δεν θα πρέπει να καταστήσουμε το καλύτερο εχθρό του καλού. Αυτό, αναφέρεται και, αυτό αναφέρθηκε και από την κυρία Μαγκάβαν. Πράγματι θα μπορούσαμε να στοχεύσουμε σε ένα εξαιρετικό πακέτο, αλλά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Το backloading θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι θα πρέπει εμείς από την 1η Ιανουαρίου του 2013 θα πρέπει να σταματήσουμε να πλημμυρίζουμε την αγορά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της αγοράς αυτής και θα πρέπει να προσπαθήσουμε τα δικαιώματα να τα κρατήσουμε για αργότερα. Θα πρέπει εμείς ε, να μην ε, κορέσουμε ακόμα περισσότερο μια κορεσμένη αγορά. Αρκετοί από εσά εκφράστηκαν αρνητικά για την πρόταση αυτή. Αλλά έχετε συμφωνήσει με αυτή την αντίληψη σε όλα τα συστήματα της αγοράς τα οργανωμένα. Δεν πρέπει εξ αρχής να πλημμυρίζουμε μια αγορά. Και αυτό κάνει το backloading. Αυτός είναι ο στόχος του backloading. Γι' αυτό λοιπόν το backloading πολιτικά μπορείτε να το δεχτείτε. Γνωρίζω επίσης ότι και οι διαρθρωτικές επιλογές είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται για πολλές χώρες και για πολλούς από εσά με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και είναι μια απόφαση η οποία θα απαιτήσει και περισσότερο χρόνο. Γι' αυτό ξεχωρίζουμε τα πράγματα, γιατί αυτοί οι οποίοι είναι ήδη μέσα στην αγορά και λειτουργούν στην αγορά θα ήταν δίκαιο το ταχύτερο δυνατόν να γνωρίζουν είναι τι τους περιμένει στα πλαίσια της επόμενης φάσης ε, των δημοπρασιών, των πληστηριασμών, συγγνώμη. Λοιπόν, είναι πράγματα που πρέπει να ξεχωρίσουμε. Για τον κύριο Σιμάνσκι, κυρία Χιούμπνερ και άλλους. Αυτοί αναφέρθηκαν σε κάτι το οποίο μπορεί έτσι και αλλιώ να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε ότι επανειλημμένα ακολουθούμε τη λογική αυτή συστηματικά προσπαθούμε να κατησχίσουμε τις αγοράς. Όχι βέβαια. Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρη στην αρχική μου παρέμβαση. Γνωρίζουμε ότι οι προτάσεις αυτές οφείλονται σε κάποιες έκτακτες συνθήκες και επιβεβαιώνω ότι κάτι τέτοιο ε, θα εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση όπου πράγματι ισχύουν αυτές οι έκτακτες συνθήκες. Δεν ξέρω ποιος αδελφό. είπε ε, ότι έχει αμφιβολίες για αυτά τα οποία είπα. Θα ε, τα, στείλω γραπτά αυτά τα οποία είπα στην αρχική μου παρέμβαση. Είναι σαφές ότι εμείς σεβόμαστε ότι το Κοινοβούλιο είναι πρώτο αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει για την τροπολογία αυτή πριν από την υιοθέτηση ασδήποτε άλλης πρότασης. Τώρα για το αν θα οδηγηθούμε σε αύξηση των τιμών και ο κύριος Κυλακάκης εδώ αναφέρθηκε σε αυτό. Να σας υπενθυμίσω εδώ ότι όταν εμείς ε, σαν κοινοβούλιο μάλλον ε, υιοθέτησε το πακέτο για την ενέργεια το 2008 οι τιμές οι οποίες προεβλέπονται ήταν γύρω στο 30 ευρώ. Τώρα έχουμε φτάσει όπως είπε ο Πρόεδρος στα 8 και 46 σέντ, δηλαδή στο 1 τέταρτο περίπου της αρχικής εκτίμησης. Δεν μπορείτε να πείτε λοιπόν ότι η τιμή αυτή δεν αντικατοπτρίζει την ισχύουσα κρίση. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε με το backloading. Προσπαθούμε να αποφύγουμε, να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα κάτω τις τιμές. Εδώ συνδέεται το θέμα και με την οδηγία για την αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας. Και εδώ εσείς σαν κοινοβούλιο είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το αντιμετωπίσει το θέμα αυτό σαν τμήμα της οδηγίας για την αποδοτικότητα της ενέργειας. Αν πάρετε χίλιες μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και αρχίσετε να επενδύετε στην αποδοτικότητα της ενέργειας όπως θα θέλατε να κάνουν, Ποια θα είναι η άμεση συνέπεια. Άμεση συνέπεια θα είναι ότι οι εταιρείε οι οποίες δεν κάνουν τίποτα θα έχουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Γιατί κάποιοι άλλοι επενδύουν στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα έχουν λιγότερα κέρδη, αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν οι τιμές και αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα θα πληρώνουν τα λιγότερα. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε να, να, να πετύχουμε. Και όσοι το συνδέεται αυτό την πρότασή μας και με την ανάπτυξη και με, με την απασχόληση, μα αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε τη συγκεκριμένη πρόταση, γιατί είναι μοχλός για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα αυτό και περί αυτού πρόκειται υποσχέθηκα να μην μακρηγορήσω. Κλείνοντας θα ήθελα να σας πω ότι ελπίζω πως το ταχύτερο δυνατόν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο ύψος ποσού και θα κατανοήσετε κι εσείς τη χρησιμότητα του backloading. Καταλαβαίνετε ότι είναι περίπλοκα τα πράγματα, είναι και περίπλοκες οι διαδικασίες και οι χρονισμοί θα έχετε την έκθεση την Τετάρτη για την αγορά του διοξιδίου του άνθρακα με όλες τις πιθανές επιλογές. Λέτε κάποιοι από εσάς γιατί δεν κάνουμε μία πρόταση και ταυτόχρονα μας λέτε να σεβαστούμε την δημοκρατία και να έχετε χρόνο για να τα συζητήσετε όλα αυτά. Αυτό θέλουν επίσης και οι εμπλεκόμενοι στις αγορές. Εμείς λοιπόν θα ορίσουμε τις επιλογές για τα πιο μακροπρόθεσμα διαφθρωτικά μέτρα. Ξέρουμε ότι η συζήτηση δεν είναι εύκολη, είναι κάτι το οποίο δεν θα λύσουμε με μια απλή κίνηση ε, ε, ε, πραγματικά δακτυλουργική. Νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε σωστότερα αυτά που ανακοινώσαμε ήδη την Άνοιξη όταν οι Υπουργοί για πρώτη φορά συζήτησαν το θέμα της αγοράς του διοξιδίου του άνθρακα όπως επίσης και του ETS. Για πρώτη φορά τον Απρίλιο είπαμε εμείς ότι θα πρέπει να ρυθμούν μέτρα μέσα στον χρόνο. Την Τετάρτη παρουσιάζουμε τα μέτρα αυτά και θα ασχοληθούμε από τη μία ειδικά με το backloading και από την άλλη με τα διαφθορτικά μακροπρόθεσμα μέτρα. Λοιπόν, ελπίζω να κατανοείτε το διακύβευμα, εν πάση Πρόεδρε, ότι το ETS μπορεί να είναι πάντα ένα ισχυρό μέσο για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα του άνθρακα όσοι γνωρίζουν την αγορά αυτή, όσοι ξέρουν να αναλύσουν την αγορά αυτή, όσοι κατανοούν τι σημαίνει η αγορά αυτή, περιμένουν πάρα πολλά από μένα, από εσά, από την Ευρώπη να πάρει μία απόφαση. Να μην ξεχνάμε ότι στην Αυστραλία θέλουν να συμφωνήσουν μαζί τους. Η Κορέα έχει κάνει το δικό της σχήμα ETS έχουμε αρχίσει και υπογράφουμε, ε, κάνουμε συζητήσεις για υπογραφή συμφωνίας και με τους Κινέζους. Η Καλιφόρνια προχωράει με το δικό της ε, και νομίζω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν και τις εξελίξεις τώρα μετά την εκλογή Ομπάμα στη ΣΥΠΑ. Λοιπόν, σκεφτείτε που βρισκόμασταν ε, πριν μερικά χρόνια ο κόσμος προσβλέπει στην Ευρώπη. Ο κόσμος υιοθετεί τους ίδιους μηχανισμούς, τους εργαζόμενους στην αγορά που εμείς απαιτείται να ενεργοποιήσουμε για να δουλέψει ακριβώς το ETS. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας τις ε, ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες, την κρίση την οποία βιώνουμε Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν είναι κάτι το απλό, αλλά θα ήταν ανεύθυνο αν σαν υπεύθυνοι δεν πάρουμε τις αποφάσεις για να δουλέψει το σύστημα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο ε, για να τα συζητήσετε αυτά. Πολλές φορές είναι πάρα πολύ τεχνικά τα θέματα, αλλά το θέμα είναι να δώσουμε τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε να δουλέψει το ETS ή μήπως όχι. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήσασταν μαζί μας σήμερα εδώ στην Επιτροπή και που μας δώσατε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας τα θέματα που προβλέπονται στο μέλλον, ή προτάσεις που έχουν δικαιωτευθεί. Σημαντικό θα είναι σε θέματα προστασίας του κλίματος να έχουμε ουσιαστικές προτάσεις, ουσιαστική συνεργασία, αξιοπιστία και για τη βιομηχανία, αλλά και για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με την ε, κλιματική αλλαγή, είναι απαραίτητο να βλέπουν ε, ένα πλαίσιο σταθερό, αξιόπιστο. Η πρόταση για το ETS και για το κλίμα έχουν κατατεθεί. Μας είπατε ότι είναι τροποποίησεις αυτέ που προτείνεται. Υπάρχουν πολλά θέματα σχετικά με το μεγάλο αριθμό των πιστοποιητικών που μας εκθέσατε και εσείς. Θα διαδραματίσουμε και θα κάνουμε και εμεί ό,τι μπορούμε από πλευρά μα. Σα ευχαριστώ λοιπόν και παρακαλώ τους ομιλητέ μας να έρθουν στο Προεδρείο για να συνεχίσουμε το δεύτερο γύρο των συζητήσεων. So, ich bitte doch alle, so langsam... Παρακαλώ να ξαναγυρίσετε στις θέσεις σας σιγά σιγά. Άπαντες.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 Και ξεκινώ με τον κύριο Χάουκε Χέρφμαν. Επιστήμονα ερευνητή στο Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Οικολογίας. Thank you very much for the invitation and the possibility. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δίνετε να συστήσουμε σας την πρόταση για το backloading. Όπως γνωρίζετε, το στο ΕΚΟ, Ινστιτούτο για την Εφηρμοσμένη Οικολογία, είναι ανεξάρτητο Ινστιτούτο. Έχουμε κάνει δύο έρευνες ανεξάρτητες για το backloading και το ETS. Όποιος ενδιαφέρεται για πιο λεπτομερείς, για πιο λεπτομερείς στοιχεία, δεδομένου ότι μέσα 10 λεπτά δεν μπορώ να κάλυψω, να κάλυψω τα πάντα, ε, καλείται να ε, ρίξει μια ματιά στις έρευνές μας, που είναι πολύ αναλυτικές και τεκμηριωμένες και θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως σε δύο σημεία. Την ε, υπερπροσφορά που έχουμε αυτή την εποχή και κάποια στοιχεία που απορρέουν από τις έρευνες μας ως προς τις συνέπειες του backloading επί των τιμών και το, τη διαρροή άνθρακα, leakage. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχω ειδήσει τόσο καλές όσο και κακές. Οι κακέ ειδήσει είναι ότι το backloading είναι ένα μόνο βήμα, αλλά δεν αρκεί για την επίλυση τη υπερπροσφορά που έχουμε. Θα χρειαστούν διαρθρωτικά μέτρα μακροπρόθεσμα. Και οι συνέπειε επί των τιμών του backloading, τη πρόταση backloading, θα είναι πολύ περιορισμένε. Αυτό όμω θεωρείται και καλή είδηση. Φαντάζομαι από όσου ε, φρονούν πω ε, θα προξενήσει το backloading πολλά προβλήματα και δυσχέρειε στην βιομηχανία ενέργεια στο κλάδο της ενέργειας. Ας ε, θίξουμε όμως πρώτα το θέμα της υπερπροσφοράς. Το 2020 θα έχουμε 1,4 δις ακόμη υπερπροσφορά. Εφόσον επιτύχει, επιβιώσει το σύστημα ETS για την πολιτική αεροπορία. Εφόσον ξεφτεί με επιτυχία. Γιατί θα έχουμε αυτό το πλεόνασμα. Κύριος λόγος είναι η υπερπροσφορά σε, του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης, CDM, και επιπλέον μια πρόβλεψη για μείωση κατά 14, ε, κατά 14 16% του ΑΕΠ σε σχέση με τις ισχύουσες τιμές θα οδηγήσει σε μια χαμηλότερη αναγκαστικά ε, προσπάθεια για το θέμα του ETS. Η δική μας αισιοδοξία μόνο στις ανανεώσιμες πηγές μπορεί να εστιαστεί. Έχουμε θετικές προοπτικές σε σχέση με το 2008. Άρα μπορούμε να περιμένουμε πλεόνασμα για το 2023 από τις καθαρές πηγές ενέργειας ενώ το backloading δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση, εκβάθρων την κατάσταση. Άρα, οι τιμές του δεξιδιού του άνθρακα θα μειωθούν, θα φτάσουν στο μηδέν, δεδομένου ότι οι τιμές τωρινές μπορούν να εξηγηθούν μόνο από το γεγονός ότι αναμένεται το κοινό θεωρεί ότι θα είναι πολύ ψηλές στο μέλλον ή ότι μπορεί να εμφανιστεί σπάνες στο μέλλον. Τώρα για να περάσω στο backloading. Οι άδειε θα πρέπει να μετακυληθούν κατά μία δεκαετία με υψηλότερους ρυθμούς μείωσης. Αναλύουμε, πρέπει να πω στις ε, μελέτες μας, τις τάσεις από τις δημοπρατήσεις και τα σχετικά έσοδα που αναμένεται ότι θα αυξηθούν. Και όπως υπόθηκε, δεν πιστεύω ότι το ETS ε θα επιβιώσει. Σε περίπτωση της για τα επόμενα χρόνια θα βρουν άλλα μέσα δημοσιονομικά τα κράτη-μέλη να το αντικαταστήσουν, πράγμα το οποίο δεν είναι ευκταίο. Κύρια ανησυχία από την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού ETS ε ήταν το θέμα της βιομηχανίας και το carbon leakage όπως ονομάζεται, η διαρροή άνθρακα. Ο σχετικός κατάλογος είχε, σημειώνω, καταρτιστεί με πολύ συντηρητικές προβλέψεις και υπολογισμούς. Ξέρετε ότι είχε υπολογιστεί το κόστος του άνθρακα και η ένταση εμπορίου. Η ένταση εμπορίου είχε λάβει υπόψη μόνο τι 27 χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν λάμβανε υπόψη χώρε όπω η Νορβηγία και η Ισλανδία που έχουν ήδη μπει στο, στο ETS της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τη Αυστραλία που θα συνδεθεί με αυτό. Άρα η ένταση εμπορίου για πολλού τομεί θα είναι χαμηλότερη όταν έρθουμε με τα πραγματικά στοιχεία. Το κόστος του άνθρακα, από την άλλη, με βάση την τιμή των 30 ευρώ, είναι τετραπλάσιο της τρέχουσας τιμής. Άρα, με αυτούς τους υπολογισμούς βλέπουμε ότι η κατάσταση τώρα αποδεικνύει πως είναι εσφαλμένη η υπολογισμική η προβλέψη και χρειάζεται προσαρμογή. Πολλές πολιτικές έχουν εισαχθεί με στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών τάσεων με ε, ένα ελεύθερο ποσοστό 1%, ένα δωρεάν ποσοστό που έχει χορηγηθεί, με διαφορετικές τιμές με ευνοϊκότερη μεταχείριση για τον βιομηχανικό τομέα στη δεύτερη φάση και τη δυνατότητα του banking κατά την τρίτη φάση έτσι ώστε να αξιοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα ορισμένε άδειε. Το backloading δεν αλλάζει αυτό το πρόβλημα της ε, ε, υπερπροσφοράς. Όσον αφορά τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, όπως λέγω, προβλήματα δεν προβλέπονται. Αλλά ως προς το carbon leakage ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα επειδή έχουμε πολύ χαμηλές τιμές και διαφορετική πυκνότητα, εμπορική πυκνότητα ή αγοράς από ό,τι αρχικά προβλεφθεί. Άρα, σπάνια για την επόμενη δεκαετία δεν προβλέπεται, το backloading δεν αρκεί, διαρθρωτικά μέτρα χρειάζονται. Χρειάζεται να ληφθούν και αυτά και αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Δεν προβλέπεται να έχει το backloading. Αυτές είναι οι δικές μας εκτιμήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χέρμαν για την παρουσίαση. Ευχαριστώ για την ομιλία σας. Ο κύριος... Η κυρία Helen Bray, ε, σύμβουλος για κλιματική πολιτική της Shell. Έχετε το λόγο. Good Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να συζητήσουμε το ETS. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι το θετικό μήνυμα το οποίο στέλνει η Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο και σε σχέση με την πρόταση για το backloading και για τον ρόλο του ETS e στην ενεργειακή πολιτική και την κλιματολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020. Στην Ευρώπη χρησιμοποιούμε και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τα χρησιμοποιούμε για την βιομηχανία, για την θέρμανση και για τις μεταφορές. Το κέντρο έρευνας και καινοτομίας ε, χρησιμοποιούν την τεχνολογία του αύριο και με βιοκαύσιμα και με την χρήση των συγκρατούμενων ποσοτήτων διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είμαστε μια ιδιαίτερα ε, ευαίσθητη επιχείρηση εκτεθειμένη στο διεθνή ανταγωνισμό. Κάνουμε προσπάθειες για να αναπτύξουμε ε, τεχνολογίες χαμηλής χρήσης άνθρακα, ε, περιορίζοντας και μετριάζοντας τις αρνητικές συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών. Ε, το θέμα της διαρροής ποσοτήτων είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και στα πλαίσια της πολιτικής μας πέραν από το 2020 πρέπει να πάρουμε μέτρα ήδη από σήμερα. Η υποστήριξη του ETS βασίζεται στις αρχές μας. Προσπαθούμε να μειώσουμε επίσης και την εκπομπή διοξίδιου του άνθρακα από τις βιομηχανικές μονάδες και από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας πρέπει φυσικά να υπάρξει μια τιμολόγηση των συγκεκριμένων αυτών εκπομπών. Πρώτον, το ανώτατο όριο εκπομπών είναι κάτι το οποίο περιβαλλοντικά θα λειτουργήσει θετικά και οδηγεί τις χώρες να μειώσουν. Το σύστημα εμπορίας μειώνει ακριβώς τις ε, ε, εκπομπές όπως το αναγνωρίζουν οι διεθνείς υπηρεσίες ενέργειας η καινοτομία και η ανάπτυξη επιτρέπουν τις αναπτύξεις ανανεώσιμων πηγών όπως επίσης και αποθήκευσης ποσοτήτων διοξιδίου του άνθρακα και η ανταλλαγή δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την προώθηση των ιδίων αυτών μορφών ενέργειας. Και μέσω ακριβώς των διεθνών δικαιωμάτων αυτών υποστηρίζουμε τη μεταφορά τεχνολογιών και προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για αυτούς τους λόγους υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το σύστημα εκπομπής το οποίο χρήζει ενίσχυσης. Όπως υπόθηκε ε, πριν, το θέμα αυτό ε, έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες, όπως Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Καναδά, τμήματα της Κίνας, Ηνωμένε Πολιτείε εν μέρη. Αυτά είναι πολύ σημαντικά βήματα για την δημιουργία μιας σφαιρικής παγκόσμιας αντιμετώπισης του σαν, χημικός, σαν χημική βιομηχανία και πετρελαϊκή βιομηχανία τα σχήματα ανταλλαγής δικαιωμάτων για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι ποσοστώσεις τις οποίες παίρνουμε βασίζονται στις βέλτιστες δυνατές τεχνολογίες, αυτές χρησιμοποιούμε προστατεύοντας και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εξαγωγές προς χώρες οι οποίες ε, δεν συμμετέχουν στην λειτουργία του σχήματος. Αυτό είναι κάτι που δίδει κίνητρα στο να είμαστε αποδοτικοί ενεργειακά και να επενδύουμε σε συστήματα χαμηλής παραγωγής διοξιδίου του άνθρακα. Είμαστε πρωτοπόροι στον κόσμο και αυτό το βοηθά ακριβώς η ύπαρξη του ETS. Τώρα για το 2020 η αγορά διοξιδίου του άνθρακα θα δώσει επιπλέον κίνητρα σε επενδύσεις στον τομέα της χρήσης ε, ε, χαμηλών εκπομπών και ανανεώσιμων πηγών. Απαιτείται ένα σταθερό πλαίσιο νομικό για το 2030. Θέλουμε συγκεκριμένους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης ε, των εκπομπών και ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε είναι μέσω ακριβώς του συστήματος ETS. Πρέπει να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα το σύστημα αφαιρώντας ένα δις δικαιωμάτων και θα πρέπει επίσης τα μέτρα αυτά σε συνδυασμό με τον καθορισμό των στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας το 2030 θα μας διευκολύνει στη χρήση νέων τεχνολογιών χαμηλής χρήσης άνθρακα. Ε, θα πρέπει ταυτόχρονα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να τονώσει τους ε, τομείς τους βιομηχανικούς και την παραγωγή ενέργειας προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί έχει σημασία και σήμερα το σχέδιο αυτό. Είναι σαφές ότι το σύστημα αυτό δεν είναι κάτι το προσωρινό είναι κάτι το που λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι μια στροφή στην οικονομική δραστηριότητα και είναι κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει πάρα πολύ στη μείωση ε, των εκπομπών σε αυτή τη δεκαετία αλλά είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να οδηγήσει στη μείωση του κόστους ε, των δικαιωμάτων που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών όπως επίσης και αποθήκευση ποσοτήτων διοξιδίου του άνθρακα. Ε, πρόκειται για μια μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών. Διαρθρωτικό κομμάτι της ε, πολιτικής της ευρύτερης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τον περιορισμό των κλιματολογικών συνεπειών. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να προκαλέσει κάποιες διαφοροποιήσεις ε, ανάμεσα στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Ο καθορισμός των τιμών ηλεκτρισμού όμως είναι κάτι το πάρα πολύ περίπλοκο όπως ε, και ε, ο μέσος όρος της τιμής του ηλεκτρισμού τον προηγούμενο χρόνο σε διάφορες χώρες της Ευρώπης κυμαίνεται από 33 σε 75 από την φθηνότερη στην ακριβότερη χώρα η τιμολόγηση ανα, ανα ώρα είναι θα έλεγα από ένα σε δύο και αυτό είναι κάτι το οποίο προκαλεί προβλήματα στους υπολογισμούς. Απαιτείται λοιπόν να προσαρμοστούμε στις έκτακτες αυτές οι οικονομικές συνθήκες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ήδη από το 2008 και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις απαιτούμενες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι πληστηριασμοί ποσοτήτων, κάτι το οποίο θα μας δώσει χρόνο για να βρούμε και τα σωστά μακροπρόθεσμα μέτρα. Λοιπόν, συμπερασματικά, πρώτον, απαιτείται ένα σταθερό πλαίσιο για το 2030 που να περιλαμβάνει ένα μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης εκπομπών. Οι επικαλεπτόμενες πολιτικές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά για να αποφύγουμε αντιτιθέμενους στόχους είναι ένα σωστός τρόπος για τη μείωση των εκπομπών στον τομέα της παραγωγής ενέργειας και στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και θα βοηθήσει την ανάκτηση κατα... ανταγωνιστικότητας και την καταπολέμηση των νεκροών ποσοτήτων διοξιδίου του άνθρακα και ακριβώς το backloading είναι κάτι που θα μας οδηγήσει στις αρχές της φάσης 3. Είναι ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα που θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία του ETS. Και αυτό θα συνδυάσει και το υπάρχον σημερινό ευρωπαϊκό patchwork μείωσης εκπομπών. Θα πρέπει εδώ να αναγνωρίσω την ηγέτιδα θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Ακολουθεί ο κύριος ε, Πέτερ Μπότσακ, ο οποίος είναι διευθυντής για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στο ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικών Βιομηχανιών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να έρθω. Και δεν μιλάω μονάχα για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χημικών Βιομηχανών, αλλά και για τη Συμμαχία Βιομηχανιών Έντασης Ενέργειας. Επομένως μιλάω και για την ιαλουργία, τη χαλιβουργία και για πολλές άλλες βιομηχανίες που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την πρόταση της Κομισιόν. Και όταν λέω ενδιαφέρονται εννοώ ανησυχούν. Ανησυχούν γιατί είμαστε ενεργοβόρες βιομηχανίες. Παράγουμε πράγματα στην Ευρώπη, αγαθά στην Ευρώπη. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό χωρίς ενέργεια. Γι' αυτό οι βιομηχανικοί αυτοί τομεί τους οποίους εγώ εκπροσωπώ ανησυχούν τα μάλα. Γιατί για μας οι τιμές έχουν μεγάλη σημασία, η αξιοπιστία και η <clears throat> ανθεκτικότητα του συστήματος είναι σημαντικές. Το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε από κοινού τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακος μέχρι το 2050 με έναν τρόπο που θα είναι ισοδίκαιος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να το πετύχουμε με το πιο αποδοτικό και το, πιο, και το λιγότερο ε, πολυδάπανο τρόπο που γίνεται. Και αυτός είναι και ο στόχος του συστήματος ETS, να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, δηλαδή μείωση των εκπομπών κατά 20%, αύξηση της αποδοτικότητας κατά 20% και επίτευξη μεριδίου ανανεώσιμων ενεργειών κατά 20%. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα εμπορίας εκπομπών λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύψει τις εκπομπές από βιομηχανικές δραστηριότητες. Δεν μιλάμε για τις εκπομπές των νοικοκυριών ή τις εκπομπές από μέσα μεταφοράς. Σήμερα <clears throat> μπορούμε να μιλήσουμε για τους τομείς που καλύπτονται από το σύστημα ETS. Και φαίνεται ότι η πορεία τους για να μειωθούν κατά 20% εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2020 είναι σωστή για τον τομέα της χημικής βιομηχανίας. Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά. Σε σχέση με το 1990 φαίνεται ότι εμείς <clears throat> μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές μας κατά 50 με 60% μέχρι το 2020. Αλλά παράλληλα είναι απογοητευτικό να βλέπουμε ότι αυτές οι βελτιώσεις, το κέρδος αυτό στις εκπομπές έχει αντισταθμιστεί από την αύξηση των εκπομπών σε άλλους τομείς. Φυσικά, φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τιμωρήσουμε αυτούς οι οποίοι επιτυγχάνουν τους στόχους επιβάλλοντάς τους υψηλότερο κόστος και υψηλότερες τιμές. Και να γίνουμε έτσι θύματα της ίδιας μας επιτυχίας. Θέλουμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών δεν είναι το μοναδικό, ούτε καν το κύριο εργαλείο το οποίο παροτρύνει για επενδύσεις σε καινοτομία που έχει χαμηλή χρυσή άνθρακα. Οι επενδύσεις βασίζονται σε τιμολόγηση η οποία δίνει στους επενδυτές τη σωστή απόδοση της επενδύσεις τους. Θεωρούνται ότι είναι επιδοτήσεις αυτές οι επιδοτούμενες τιμολογίες, αλλά τελικά το κόστος τους το επομίζεται ο τελικός καταναλωτής, ο φορολογούμενος. Για την πρόταση του backloading. Πιστεύουμε ότι πολλές από τις εξοικονομήσεις χρήσης ενέργειας μέχρι στιγμή ήταν αποτέλεσμα της τιμολόγηση ενέργειας, των τιμών ενέργειας. Αυτή όμως τη χρονική στιγμή οι εταιρείε μας πληρώνουν μέχρι πέντε φορές μεγαλύτερη τιμή για το φυσικό αέριο στην ε, Ευρώπη από ότι οι Αμερικάνοι ομολογοί μας. Ποιο λοιπόν δεν θα ήθελε να κάνει εξοικονόμηση ενέργειας στο βαθμό του δυνατού. Το γεγονός επίσης ότι άλλοι τομείς που δεν υπόκεινται στο σύστημα εμπορίας δεν προχωρούν σε μειώσεις αλλά αυξάνει τις εκπομπές, αυξάνει εκπομπές τους μπορεί να υποσκάψει τις προσπαθίες μας. Είναι σαφές ότι το set aside και οι υψηλέ τιμές για τον άνθρακα δεν θα λύσουν το πρόβλημα αυτό. Όταν παρουσιάζεται εκτός του συστήματος εμπορίας, επίσης και το σύστημα ETS δεν παροτρύνει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες ενέργειες και το backloading, ούτε και αυτό θα οδηγήσει σε επενδύσεις προς την κατεύθυνση αυτή, ακόμα και αν πολλοί θα το έλπιζαν αυτό. Επομένως είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς πως το backloading και το set aside μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω και ταχύτερες μειώσεις στις εκπομπές διοξιδίων του άνθρακος. Ενδεχομένως δεν είναι καν η πρόθεση της πρότασης της Κομισιόν να γίνει κάτι τέτοιο. Ίσως η πρόταση της Κομισιόν είναι να δώσει περισσότερα έσοδα στις κυβερνήσεις. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ρωτήσουμε αν αυτό θα γίνει γεγονό. Αν ατενίσουμε τους εμπλεκόμενους που υποστηρίζουν το backloading και το set aside, πρόκειται για ένα συνασπισμό συμφερόντων ουσιαστικά. Αν δούμε ποιοι βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα, θα πρέπει να πω καταρχήν ότι εμείς ως ενεργοβόρες βιομηχανείς υποστηρίζουμε το ETS γιατί είναι ένα κομβικό εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών. Αυτό όμως το οποίο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε είναι να μετατραπεί το ETS σε ένα εργαλείο που μπορεί να άρει άλλους υποστηρικτικούς μηχανισμούς. Γι' αυτό ανησυχούμε ότι υπάρχει πληθώρα ίσως και υπερβολική πολυπλοκότητα στα εργαλεία αν ακολουθήσουμε τη νέα πρόταση της Κομισιόν και θα θέλαμε να ξέρουμε πότε τελικά θα είναι ικανοποιημένοι με την τιμή του άνθρακος οι νομοθέτες και ποιος είναι ο αντικειμενικός του στόχος. Πιστεύουμε ότι η αύξηση της τιμής του άνθρακα δεν θα οδηγήσει σε επενδύσεις σε τεχνολογία χαμηλής χρήσης άνθρακα, ιδίως όταν βρισκόμαστε σε μια τόσο βαθιά οικονομική κρίση αν δω του, τα αριθμητικά στοιχεία, το Σεπτέμβριο η Ευρώπη έχει χάσει μόνο το Σεπτέμβριο 170.000 θέσεις απασχόλησης. Είναι λοιπόν πολύ υψηλή αυτή η απώλεια. Όταν χάνουμε 100.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πολιτικές οι οποίες θα προωθήσουν τις τιμές της ενέργειας και με τον τρόπο αυτό να βοηθήσουμε τις επενδύσεις. Αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε επίσης <clears throat> είναι ότι η παραγωγή ηλεκτρισμής ενέργειας είναι σε θέση να μετακυλίουν πάντα το πρόσθετο κόστος. Και το αποτέλεσμα τελικά για μας είναι ότι αυξάνει ο πληθωρισμός ενώ αυτοί οι οποίοι παράγουν ενέργεια από τον άνθρακα εξακολουθούν να είναι κερδοφόροι γιατί μπορούν πάντα να μετακυλήσουν το κόστος στους ε, καταναλωτές ενέργειας. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο σημείο εκκίνησης. Δεν υπάρχει κάποιο πρόσθετο κίνητρο για να υπάρξουν επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες ή σε τεχνολογίες χαμηλής χρήσης άνθρακα. Αυτό το είδαμε και από το παρελθόν όταν είχαμε δώσει στους παραγωγούς ενέργειας δυνατότητα να κάνουν ε, τεράστια κέρδη και περιμέναμε να επενδύουν αυτά τα κέρδη σε τεχνολογίες χαμηλής χρήσης άνθρακα ή σε καθαρότερες τεχνολογίες. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτές οι επενδύσεις πράγματι θα λάβουν χώρα. Απλώς έχουμε εξασφαλίσει την αύξηση των τιμών ενέργειας. Επομένως, εν κατακλείδη, Εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα με το οποίο δίνουμε, μεταφέρουμε τον πλούτο από τα νοικοκυριά και από τους χρήστες ενέργειας σε κάποιους ενδιαφερομένους κύκλους και τομείς. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε το ερώτημα. Αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερα έσοδα για τις κυβερνήσεις. Αναρωτιόμαστε, έχουμε αμφιβολίες γιατί βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός θα ε, μειώσει την οικονομική δραστηριότητα και θα οδηγηθούμε σε μια διπλή ύφεση. Επομένως ανησυχούμε για όλες αυτές τις ιδέες. Αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγουμε αυτή τη στιγμή είναι οποιοδήποτε μέτρο το οποίο θα εδραιώσει την κατάσταση ύφεση στην οποία βρισκόμαστε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι, και εδώ υπήρξε και ένα ερώτημα που είχε διατυπωθεί από τη Λίντα Μακίουαν προηγουμένω. Πολύ καλά. Τι προτείνετε λοιπόν, αν δεν θέλετε μια τέτοια αντιμετώπιση λέμε, εμείς βλέπουμε να υπάρχουν ψεγάδια στο ETS, δεν είναι τέλειο σύστημα. Αλλά δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή που θα πρέπει να παρέμβουμε στο σύστημα αυτό. Μετά από το 2020 και μόνο πρέπει να παρέμβουμε. Θα πρέπει τώρα να σκεφτούμε για τις προτάσεις που αφορούν την τέταρτη περίοδο για το ETS τότε θα ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι και μπορούμε να διδαχτούμε από τα τωρινά σφάλματα του περιβάλλοντος. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν πολλά συμφέροντα στην Κίνα, στην Καλιφόρνια, στην Αυστραλία που ήδη έχουν μάθει από τα, από τα λάθη μας και που θα, όλοι αυτοί θα σχεδιάσουν ένα τελείως διαφορετικό σύστημα από αυτό που ισχύει στην Ευρώπη. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να μάθουμε να, από τους άλλους και από τα δικά μας φάρματα και να υπάρξει μια μεγαλύτερη σύγκληση προσπαθειών και εδώ θέλουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο, ένα ενεργό ρόλο για να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα αλλά και για να διευκολύνουμε μια αποτελεσματική μετάβαση και μια μετάβαση που θα γίνει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρος, κύριε Μπότσα. Είστε εδώ προσκεκλημένος εκπροσωπός της ΦΙΣΙΚ. Μιλάτε και εκ αυτή τη και εν τέλει, παρακαλώ τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΙΕΤΑ, International Emissions Trading Association, κύριο Dirk Φόριστερ, να λάβει το λόγο. Μετά ο κύριος Ντεβέκερ από την Γενική Διεύθυνση τα λάβει το λόγο τελευταίος. Κύριος Φόριστερ, ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ πολύ που επιτρέπετε στην ε, Διεθνή Ένωση Ανταλλαγών Εκπομπών, η ΕΤΑ, να έρθει. Ελπίζω να γνωρίζετε ποιοι είμαστε. Εκπροσωπούμε 150 εταιρείε που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ε, ανταλλαγών εκπομπών. Οι περισσότερες από τις ε, επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε ασχολούνται με τις εκπομπές ανταλλαγές εκπομπών, ενώ οι λοιπές, λιγότερο το 5%, είναι περισσότερο στο χώρο της επαλήθευσης, της επιθεώρησης εποπτείας της λειτουργίας του συστήματος. Άρα λοιπόν έχουμε κάθε ενδιαφέρον για το θέμα αυτό του ETS. Ε Η ΕΤΑ λοιπόν στηρίζει το ETS ε πάντα ως τον καλύτερο μέχρι στιγμής μηχανισμό για την επίτευξη των, της πίωσης των εκπομπών με χαμηλό κόστος και χαιρόμαστε για την εισαγωγή της ευρωπαϊκή πολιτική. Πιστεύουμε ότι η πολιτική αυτή είναι καλύτερη ανά τον κόσμο. Είχε 160 δις 126 δις σε συναλλαγές σε άνθρακα ανά τον κόσμο με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, του σύστημα ITS, ε άρα είναι πολύ καλό. Έχει προσφέρει και κατευθύνσεις ή προσανατολισμούς για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων και άρα πιστεύουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να μας επιτρέψει να επιτύχουμε έναν επιδιωκόμενο στόχο με χαμηλό κατά το δυνατό κόστος. Ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και ο στόχο προστασία του περιβάλλοντος που ασφαλώ γνωρίζετε καθώ είναι η δουλειά σα. Πιστεύουμε ότι το ETS έχει εξυπηρετήσει σημαντικά και τον στόχο της αποδέσμευσης της δημιουργικότητας του χώρου της βιομηχανίας. Πολλοί είναι οι επαγγελματίες ανά την Ευρώπη, αλλά, ιδιαίτερα, αλλά γενικότερα και ανά τον κόσμο, που εργάζονται και βρίσκουν νέες ιδέες και σχέδια για την ε, μείωση των εκπομπών. Και έτσι παρά τις δύσκολες εποχές που ζούμε, είναι το ETS ε πρότυπο για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Στην Αυστραλία, την οποία πρόσφατα ε, επεσκέφθην εκφράζεται μεγάλη υποστήριξη για το σύστημα αυτό του, της, το ευρωπαϊκό ETS. Η Καλιφόρνια, το Κεμπέκ, οι βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, ε, πολλοί άλλοι εταίροι αναπτύσσουν προγράμματα για ανταλλαγές εκπομπών ελπίζοντας ε, κάποια μέρα να μπορέσουν να τα συνδέσουν με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι κύριες εξελίξεις σημαίνονται αυτή την εποχή στην Κίνα, πρέπει να πω, όπου πολλές ε, είναι οι επαρχίες αυτή τη στιγμή οι οποίες προσπαθούν να αναπτύξουν τα δικά τους ETS, ε ελπίζοντας, προσβλέποντας κάποια στιγμή να τα συνδέσουν με το ETS ε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ETS ε επίσης έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας βιομηχανίας πλαισίου με 4.000 τουλάχιστον έργα ε, που οδηγούν, που συζητούν για τη μείωση, που επιδιώκουν τη μείωση των ε, εκπομπών και ταυτόχρονα άλλοι 4.000 ε, που πλαισιώνουν τις προσπάθειες. Έχουμε ειδικού επαγγελματίες ανά τον κόσμο εξειδικευμένους στην μείωση των εκπομπών και στη λειτουργία της σχετικής αγοράς. Το ενδιαφέρον της Κίνας για το μέσο αυτό ανταλλαγών γεννάται και οφείλεται ακριβώς στην επιτυχία του ETS. Πάντως και παρά τις αλλαγές αντιμετωπίζει μια από τις κύριες ε, από τις μεγαλύτερες δυσκολίες της ιστορίας του το ETS, λόγω των γενικότερων συνθηκών που εξετέθησα, μετά την ε, ύφεση και την οικονομική κρίση που διαπιστώνεται, μειώνεται η λειτουργία του ETS, ε, πέφτουν ραγδαία οι τιμές και πέραν του πλήγματος που υφίστανται από τις χαμηλές τιμές οι επιχειρήσεις, δυσκολεύει το πεδίο και ως προς τις επενδύσεις. Και άρα είναι δύσκολο να κάνουν τον προγραμματισμό τους, πράγμα το οποίο με τη σειρά του ε, δυσκολεύει τις συνθήκες του ETS, ε, επιδεινώνει τις συνθήκες, οδηγεί σε στρέβλωση των τιμών και άρα θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεταρρυθμίσεις για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα, γιατί θέλουμε το ETS να παραμείνει το κύριο εργαλείο για την πολιτική και το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό η ΕΤΑ υποστηρίζει το backloading σαν ένα βραχυπρόθεσμο μέσον που όμως θεωρούμε ότι θα είναι αποτελεσματικό μόνο αν το ακολουθήσει, το συνοδεύσει και μια σειρά από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέγει ότι θα είναι ένα στιγμιαίο και βραχυπρόθεσμο ε, μέτρο έτσι ώστε να κερδίσουμε χρόνο για την γενικότερη συζήτηση που αφορά τις διαφορετικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Ως προς τα ποσά, τι ποσότητες που θα πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα του backloading δεν τοποθετούμεθα. Απλώ πιστεύουμε ότι είναι μια καλή λύση γενικά. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράσεις κατά τρόπο διαφανή και τις αποφάσεις της να τις κοινοποιεί έγκαιρα ώστε να ετοιμάζονται οι επιχειρήσεις για τις αλλαγές. Είναι απαραίτητο να μην καθυστερήσει αυτή η πρόταση να ε, προχωρήσει. Ξέρουμε ότι θα, θα δημοσιοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή το χειρότερο δυνατό. Επίσης η ΕΤΑ καλεί τους αρμόδιους για τη λήψη των αποφάσεων να προχωρήσουν σε ουσιαστικέ διαρθρωτικέ αλλαγέ. Και ενώ γνωρίζουμε ότι μόλι έχει ξεκινήσει η συζήτηση, θα θέλαμε να υποβάλουμε κάποιε ιδέε για σκέψη. Έχουμε κάνει μια ανάλυση τεσσάρων διαφορετικών εναλλακτικών ως προς τις διαφορετικές με, μεταρρυθμίσεις και, εδώ, και δεν έχουμε κάποια επιλογή προτίμησης προς το παρόν, πιστεύουμε ότι θα ήταν καλό να έχουμε τη δυνατότητα για μια διεξοδική ανταλλαγή απόψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας να δούμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να υποστηρίξουμε ιδέες και να προσφέρουμε την ε, ενθάρρυνσή μας στις προτάσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια μακροπρόθεσμη λύση ε, περνώντας πρώτα από την διαδικασία του backloading. Αν και πρέπει να πούμε ότι οι διασωτικές μεταρρυθμίσεις ίσως χρειαστούν πολύ περισσότερη προσπάθεια και πειθό το backloading πρέπει να προχωρήσει. Ωστόσο νομίζω ότι είναι ο σωστό δρόμο, και θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, καταληκτικές παρατηρήσεις ότι θα πρέπει όχι μόνο να δούμε το backloading σαν ένα μέσο ε, ανάκαμψης βραχυπρόθεσμης, αλλά και ω έναν τρόπο να πείσουμε τι αγορέ, ότι το ETS είναι μακροπρόθεσμα το σωστό μέσο και ο μηχανισμό, έτσι ώστε να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη των αγορών στο μηχανισμό. Ωστόσο αυτό ταυτόχρονα θα πρέπει να διευκρινιστεί το πώ θα γίνει, δηλαδή ώστε να μην δοθεί καμία εντύπωση στι αγορέ, ότι θα γίνεται backloading κατά καιρού τακτικά. Πρέπει λοιπόν την παρέμβαση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την ελέγξει με πολύ μεγάλη προσοχή. Και δεδομένου ότι εγώ ε, έχω συνεργαστεί στο σχεδιασμό του UETS ο σύμβουλο, σύμβουλος αλλά και στο θέμα των ε, σχετικών προγραμμάτων για τι εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα στι ΗΠΑ, μπορώ να είμαι σε θέση να σα ε, πω ότι ο χρυσό κανόν είναι πάντοτε να ορίζει κανείς τους όρους του παιχνιδιού και να αφήνει την αγορά να λειτουργεί μόνη της και ανεξάρτητα. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε μια κρίσιμη καμπή όπου χρειάζεται μια μικρή τροποποίηση του χρυσού κανόνα με αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα είναι η μόνη όμως, πρέπει να είναι η μόνη παρέμβαση να γίνει, να γίνει και σε συνεννόηση με τις επιχειρήσεις και με μια έγκαιρη προειδοποίηση, ενημέρωση ώστε να μην ε, ε, εμφανιστούν κλειδονισμοί στις αγορές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον Γιώζεφ Μπέκερ, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της ε, για την Κλιματική Αλλαγή. Για την άποψη τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να σημειώσω τρία σημεία. Όλοι θα συμφωνήσουμε καταρχά ότι το ETS τεχνικά εργάζεται και εργάζεται πολύ καλύτερα με αυτά τα οποία γινόντουσαν στο παρελθόν. Εκεί όπου δεν πάει καλά είναι γιατί δεν καταφέρνει να στείλει ένα μήνυμα στην αγορά για επενδύσεις στον τομέα των χαμηλών εκπομπών. Και δεν διευκρινίζει ακριβώς το τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο καινοτομίας με τις παρούσες χαμηλές τιμές. Ε, για πάνω από μία δεκαετία η μείωση της χρήσης του άνθρακα ήταν δεδομένη, αλλά από το τελευταίο χρόνο αυξάνεται η χρήση του άνθρακα. Βλέπουμε για πρώτη φορά λοιπόν μετά από 10 χρόνια κάποιες νέες αποφάσεις να λαμβάνονται και να δημιουργούνται νέοι εξοπλισμοί και νέες μονάδες παραγωγής ε, ενέργειας από άνθρακα. Και αυτό είναι ακριβώς απόδειξη του λάθος δρόμου τον οποίο ακολουθούμε και οι εμπλεκόμενοι λέγουν ότι με την πολύ χαμηλή τιμή και με τις χαμηλές σχετικές τιμές του άνθρακα η απόφαση αυτή είναι λογική. Εκεί ακριβώς θα θέλαμε να υπάρξει μια διαφορετική λύση. Το δεύτερο, ε, η δεύτερη παρατήρηση σχετικά με, αυτά που είπε ο Συμφωνούμε ότι στον τομέα της απασχόλησης αυτό το οποίο έχει σημασία σε τομείς όπως η χαλιβουργία, η τα τσιμέντα, η ναυπηγοεπισκευαστική είναι θα έλεγα κομβικές ε, κομβική κλάδη για τις χαμηλές εκπομπές και δεν θα δούμε αύξηση της απασχόλησης. Εκεί δεν βλέπουμε αύξηση της απασχόλησης, βλέπουμε αύξηση της ανεργίας. Και όταν ε, υποθέτουμε ότι θα πρέπει να πετύχουμε υψηλότερες τιμές, αυτό σημαίνει ότι δεν φταίνε για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα οι υψηλές τιμές. Υπάρχουν διότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες όπως ακριβώς ε, το, η παραγωγή φυσικού αερίου από σχιστολίθους στις Ηνωμένε Πολιτείες κτλ. Αυτό το οποίο θέλουμε να αποδείξουμε λοιπόν είναι ότι η ανταγωνιστικότητα με τις υπάρχουσες τιμές, με τις ισχύουσες τιμές δεν είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να ε, συνδεθεί και το ίδιο αφορά και τη σύνδεση των υψηλών τιμών με την παρούσα κατάσταση. Τώρα για μια ε, παρατήρηση της Επιτροπής. Η πρόταση της Επιτροπής για το backloading δεν ασχολείται με το περίσευμα δικαιωμάτων που έχει σωρευθεί από, την, από τις επιχειρήσεις. Εμείς παρακρατούμε θα έλεγα κάποια δικαιώματα τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να δημοπρατηθούν, ανήκουν στις δημόσιες αρχές θα έλεγα, αλλά δεν δίδονται δωρεάν και ό,τι έχει δοθεί δωρεάν ε, παραμένει δωρεάν. Γνωρίζουμε ακριβώς ότι ε, ε, δικαιώματα έχουν σωρεύσει οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και αν οι τιμές αυξηθούν φυσικά και η αξία αυτών των αποθεμάτων θα αυξηθεί κάτι το οποίο θα είναι πολύ θετικό για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Τέλος θα ήθελα να κάνω μια προκαταρκτική ανακοίνωση μετά από αυτά που είπε και η συνάλφος Χέδεγκάρτ. Σήμερα στις 8 το βράδυ το ποσό το προτινόμενο για backloading θα δημοσιοποιηθεί. Έχει ήδη προανακοινωθεί σε επίπεδο διαδικτύου και από τις 8 20 ε, ώρα απογευματινή εν πάση περιπτώσει θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση ε, της ποσότητας των δικαιωμάτων τα οποία ε, προορίζονται για backloading. Ευχαριστούμε. Με μεγάλη χαρά θα πληροφορηθούμε λοιπόν για τα ποσά αυτά που θα ανακοινώσει η Κομισιόν. Και τώρα ανοίγω τον γύρο παρεμβάσεων των συναδέλφων. Καταρχήν ο Μπάς Άουκχαουτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα στον κύριο Χέρμαν και στον κύριο Μπότσακ. Για τον κύριο Χέρμαν. Το κάνατε σαφές ότι αυτή τη στιγμή η τιμή του άνθρακα στο σύστημα ETS ε βασίζεται μονάχα σε κερδοσκοπικές συναλλαγές. Τι θα γίνει με την τιμή αυτή που τώρα βασίζεται στην κερδοσκοπία των εμπορευμένων εάν δεν εφαρμοστεί η πρόταση για το backloading. Πού θα πάει η τιμή του άνθρακος, του διοξιδίου του άνθρακος, κατά την άποψή σας. Γιατί πολλοί διαμαρτύρονται για ψηλές τιμές, ότι θα ανέβουν οι τιμές. Τι θα γίνει λοιπόν εάν είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα κερδοσκοπία στο η αρχή. Δεύτερον, για τα διαρθρωτικά μέτρα, είπατε πολύ σαφώ θέλουμε τέτοια διαρθρωτικά μέτρα. Κατά την άποψή σα, τι είναι αυτό το οποίο δίνει το πιο σαφέ μήνυμα στι αγορέ για τα διαρθρωτικά μέτρα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν έξι τέτοια μέτρα που θα προτείνει η Κομισιόν. Ποιο από τα έξι θα δώσει το καλύτερο μήνυμα στι αγορέ. Για τον κύριο Μπότσακ. Σα ευχαριστώ που μιλήσατε εξ των χρονοβόρων βιομηχανιών, των ενεργοβόρων μάλλον βιομηχανιών. Τι θα κάνουν όμως οι χαλιβουργοί και οι τσιμεντάδες, οι λεγόμενες fat cats, ευτραφείς γάτες που καταλαλώνουν μεγάλη ενέργεια, τι θα κάνουν με τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν σώρευσει. Ξέρουμε ότι αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τη μεγαλύτερη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος. Επίσης είπατε ότι υποστηρίζετε τον μακροχρόνιο, μακροχρόνιου στόχους, αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ακολουθούμε ένα δρόμο που είναι αποτελεσματικός σε επίπεδο αφόλειας, ωφέλειας σε σχέση με το κόστος για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Θεωρούμε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει το 2020 να έχουμε μια μείωση κατά 25% στην κατανάλωση ενέργειας. Τι θα γίνει λοιπόν αν δεν υπάρξει προσαρμογή στο ETS, πώς θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Τρίτο ερώτημα. Από τους οδικούς χάρτες, παραγωγός χάρη για τη χαρτοβιομηχανία, χρειάζεται να υπάρξει μια τομή στις τεχνολογίες τους, ώστε μακροχρόνια να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Για να υπάρξουν τέτοιε τεχνολογίες χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζονται χρήματα. Αλλά ξέρουμε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα του ETS για αυτές τις ε, τεχνολογίες. Με το τωρινό σύστημα δεν θα υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησης για αυτές τις τεχνολογίες, οπότε θα παραμείνουν τα προβλήματα για μακροπρόθεσμα. Τι θα γίνει με αυτό. Τέταρτο ερώτημα. Εφόσον σας ενδιαφέρουν οι στεναρές και ανθεκτικές πολιτικές, δεν θέλετε κάποιες προσαρμογές στο backloading, θα κρατήσετε την τωρινή πολιτική αλλά τότε φαίνεται ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τον κατάλογο για τη διαρροή άνθρακα, για τις μετεγκαταστάσεις που βασίζονται αυτή τη στιγμή σε μια τιμή διοξιδίου του άνθρακος που είναι 30 ευρώ. Ίσως λοιπόν πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτόν τον κατάλογο για τη διαρροή άνθρακος, ο οποίος βασίζεται στην πραγματική τιμή του άνθρακα και που εξαρτάται και από τις πολιτικές που ακολουθούνται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελβετία, Κορέα, Νορβηγία, Νότια Αφρική κτλ. Και ελπίζω ότι και εσείς προσβλέπετε σε μια μεταρρύθμιση αυτού του κανόνα γιατί αν δεν γίνει το backloading θα πρέπει να αλλάξουμε και αυτό τον κατάλογο. Έχετε κάποια απάντηση γι' αυτό. Ευχαριστώ Μπάς. Η Ρωμάνα Γιόρνταν τώρα. Σας ευχαριστώ. Ο πολιτικός στόχος του ETS είναι η μείωση των εκπομπών. Αυτός ο πολιτικός στόχος όμως δεν είναι το να ελέγχουμε τους μηχανισμούς της αγοράς. Δεν είναι να καθορίζουμε την ιδανική τιμή του άνθρακα. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να αποφασίσει η ίδια η αγορά. Έχω εδώ ένα ερώτημα για την κυρία Μπρέι από την Shell. Ωραία η ομιλία σας, αλλά έχει πολιτικό χαρακτήρα η ομιλία σας δεν είχατε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία να μας παρουσιάσετε. Ο κύριος Μπότσακ από την άλλη πλευρά μας έδωσε διάφορα στοιχεία, πληροφορίες και μας εξήγησε γιατί ανησυχεί για την πρόταση του backloading. Είπε ότι αυτή η πρόταση <clears throat> δεν θα φέρει κάποιο πρόσθετο βάρος για τον τομέα παραγωγής ενέργειας, γιατί μπορούν να μετακυλήσουν το κόστος της στα νοικοκυριά. Κύριε Μπρέι, να, μου πείτε το εξή. Σε ποιο βαθμό μπορείτε εσεί να μειώσετε τι εκπομπές επιπλέον, εάν εγκριθεί η πρόταση για το backloading. Δεύτερο ερώτημα. Πώς αυτή η πρόταση για το backloading θα επηρεάσει τις ε, χρηματοοικονομικές σας παραμέτρους. Τι θα γίνει αν υιοθετήσουμε ένα από τα σενάρια που θα μας προτείνει η Κομισιόν. Τι θα αλλάξει σε επίπεδο χρηματοοικονομικό για σας. Κυρία Χίμπνερ. Θα ήθελα να σταθώ κυρίως στην παρέμβαση του κυρίου Χέρμαν και να θέσω τις εξής ερωτήσεις. Καταρχάς, θα συμφωνούσατε ότι η αύξηση της προσφοράς στον τομέα ε, των, της, ε, ε, των εκπομπών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να μην πλημμυρίσει η αγορά. Αυτό πώς θα το οργανώσετε τεχνικά. Δεύτερον, μας είπατε ότι αυτές οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, ε, ιδιαίτερα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργούν προβλήματα. Τι ζητάτε όμως ακριβώς. Πιστεύετε ότι μία 20% σε σχέση ε, με το στόχο που έχουμε για το 2020 λόγω ακριβώς του συστήματος των τιμών έτσι όπως λειτουργεί σήμερα. Εμείς έχουμε θέσει κάποιους ε, φιλόδοξους στόχους. Σε τι αναφέρεστε λοιπόν όταν εσείς μιλάτε για το πεδίο εφαρμογής αυτών των αποφάσεων. Κόρχολα. Ευχαριστώ. Η ερώτηση με τον κύριο Τίλμπη μάλλον. Αλλά ξεκινώ ρωτώντας ποιο είναι τέλειο στόχος μα, να μειώσουμε τις εκπομπές ή να προστατεύσουμε ένα μέσον της πολιτικής για το κλίμα. Δεν είναι από τα μέτρα που έχουμε στη θέση μας. Βεβαίως και θέλω να πέσουν ε, οι εκπομπές, αλλά με χαμηλό κόστος. Δεν μπορούμε να έχουμε πληθωριστικές τιμές λόγω της έλλειψης ανταγωνιστικότητας. Ο χειρότερος εχθρός του ETS εάν θέλουμε βέβαια ότι θέλουμε να το διασώσουμε, είναι η ίδια επιτροπή για μένα. Διότι δεν πιστεύει στο μηχανισμό της αγοράς. Είναι πολλά τα χρόνια που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημιουργούσε διαφορετικά μέτρα, επικαλυπτόμενα κιόλας με το ETS, που είχαν ως συνέπεια διατάραξη της λειτουργίας του. Είτε πρόκειται για επιδοτή, είτε για άλλα μέτρα, αυτά παρεμπόδισαν τη λειτουργία μιας αγοράς εκπομπών. Επομένως, αν θέλουμε να λειτουργήσει το ETS, πρέπει να το αφήσουμε να λειτουργήσει. Και μένει είναι δύσκολο να δω πώς μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες ή ταχύτερες μειώσεις στον ανθρακά η πρόταση για το backloading που τελικά μπορεί και να μην είναι ο στόχος της ε, υποβολής της πρότασης αυτής. Μπορεί να είναι απλώς ζήτημα ε, εισοδηματικό, ε, μεγαλύτερο κέρδος για τα χώρες από τις δημοπρατήσεις. Ούτε και μας λέγεται πουθενά ότι θα γίνουν επενδύσεις σε τεχνολογία χαμηλή επιβάρυνση άνθρακα. Ως εκ τούτου... θα πρέπει να καταβάλει η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια υψηλότερο τίμημα για τις εκπομπές, δεν θα υπάρχει περιθώριο για επενδύσεις σε καθαρή τεχνολογία και επιδεινώνεται κατάσταση. Γιατί λοιπόν θεωρείτε ότι βάση πρέπει να είναι οι τιμές του ETS, ε γιατί θεωρείτε ότι είναι ένδειξη αποτυχίας οι χαμηλές τιμές για τον ε, άνθρακα, γιατί δεν βλέπετε αυτό σαν μια ένδειξη ότι επιτυγχάνουμε το στόχο μας είναι χαμηλότερη η ζήτηση και μοιραία θα μειωθεί μέχρι σε εξαφανίσεις, μέχρι σε η ζήτηση για, τις, ε, για τα πιστοποιητικά άνθρακα. Αυτό δεν θέλουμε τελικά. Ο κύριος Δέβη. Εν μέρη θέμα της συζήτηση στην ακρόασή μας ε, είναι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για το ETS. Για το ETS αυτό βλέπουμε να επικρατεί ως θέμα συζήτησης. Εγώ Παρακολουθώντα τη συζήτηση βλέπω με έμφαση την επιφλεκτικότητα που επικρατεί ως προς την αντιμετώπιση παγκόσμιας ε, αναθέρμανσης του πλανήτη που διαπιστώνω να εκφράζεται μέσα από τις παρεμβάσει που ακούστηκαν. Μας λέτε λοιπόν να κάνουμε τα ρυθμίσει πριν έχουμε το περιθώριο του χρόνου ακόμη να ε, δούμε μακροπρόθεσμα τις εξελίξεις του ETS. Ε Ίσως μέχρι τότε να έχει αλλάξει το πολιτικό κλίμα Ίσως μέχρι τότε να έχουμε συνείδηση ότι είναι κατεπίγουσα η ανάγκη να προγραμματίσουμε το μέλλον μας. Εν πάση περιπτώσει, για το backloading που πιο πολύ από όλα με απασχολεί. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Θα ήθελα να μου πούν λοιπόν οι εκπρόσωποι εδώ οι ειδικοί τι προβλέψεις έχουν σαν συνέπειες του backloading σε τιμές και συνέπειες της μη εισαγωγής του συστήματος του backloading. Γιατί κάποιοι εκπρόσωποι κυβερνήσεων που με επισκέφθηκαν μου είπαν ότι δεν έχουν αντίρρηση, ότι έχουν ε, πολλέ αντίρρησει για το backloading, αλλά θεωρούν ότι είναι πιο επικίνδυνο το να μην εισαχθεί το backloading. Γιατί μπορεί να έχει πολύ δυσμενεί συνέπειε η απουσία για τι ρύθμιση. Έτσι λοιπόν, διορθώστε με ή συμπληρώστε αν τυχόν ε, έχω απατηθεί κτρά. Πολλές φορές μας λένε ότι το ETS είναι ένας μηχανισμός αγοράς, δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στην αγορά, λειτουργεί τέλεια και ούτω καθεξής. Όμως η πρόταση της Επιτροπής μας δείχνει ότι υπάρχει ένα σύστημα αδειών που θα επικρατήσει για τα επόμενα χρόνια και εγώ, Φερρυπίν, έχοντας υπόψη ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων που το 2008 παρήγαγε χίλια αυτοκίνητα την ημέρα. Μετά έπεσε η αγορά λόγω τη οικονομική κρίση και εξακολουθεί όμω παρόλα αυτά το εργοστάσιο αυτό να παράγει χίλια αυτοκίνητα την ημέρα και άλλα χίλια την επόμενη μέρα και άλλα χίλια την παραπάνω μέρα που όμω δεν μπορεί να πουλήσει και έτσι τα αποθηκεύει γύρω-γύρω στα πάρκινγκ και γύρω-γύρω στα οικόπεδα και γενικά ε, στα αγροτεμάχια και έτσι γεμίζει ο κόσμο με πολλέ χιλιάδε αυτοκίνητα παράγονται ανά χίλια την ημέρα. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να επιδιώξει το εργοστάσιο αυτό να πουλήσει τα αυτοκίνητά του για να κερδίσει ε, ε, χρήμα, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει να τα παράγει αφού έχει εκατομμύρια αυτοκίνητα πλέον παρκαρισμένα γύρω-γύρω στην ζώνη γύρω από, το, από τις εγκαταστάσεις του. Αυτό είναι το πρόβλημα του ETS λοιπόν. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι συνεχίζουμε να παράγουμε τα αυτοκίνητα χωρίς να μπορούμε να τα πουλήσουμε ε, μέχρι ότου μπορέσει να ανακάμψει η αγορά. Συμφωνείτε με αυτή την ιδέα, με αυτή την εικόνα ή θεωρείτε ότι είναι τελείως λάθος. Ο κύριος Chris Davis, ειδικό της βιομηχανιας Κυρία Μακάβεν. Η παρατήρηση περισσότερο είναι παρά ερώτηση. Ε, την επαναλαμβάνω πάντως, την ακούστηκε και νωρίτερα, για το τι συνέπειε μπορεί να έχει το να μην κάνουμε τίποτα ή, αντίστοιχα, τι συνέπειε μπορεί να έχει το, το backloading. Εάν δεν αναλάβουμε δράση για την αποκατάσταση του προγράμματος σε σχέση με το ε, σύστημα αυτό, τι κάνουμε με τις χώρες εκείνε που ήδη έχουν επενδύσει στις καθαρές τεχνολογίες. Πώς μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όταν ξέρουμε ότι οι Πολιτείες επενδύουν ήδη σε ε, καθαρή τεχνολογία στη βαριά τους βιομηχανία, όπως άλλωστε κάνει και η Κίνα. Και ξέρουμε ότι με την θέσπιση του συστήματος των τολαγόλων είχαμε πει εξ αρχής ότι χρειάζονται κίνητρα. Εάν όμως δεν κάνουμε τίποτα τώρα, τώρα ουσιαστικά φέρουμε σε δυσμενέστατη θέση της χώρας τις επιχειρήσεις αυτές, τις υπονομεύουμε ουσιαστικά. Να, επιστολές που λέτε, ο κλάδος είναι και διαιρεμένος στην υπόθεση αυτή. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που δεν το θέλουν το ETS. Ε, άλλες επιχειρήσεις έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποτελεσματικότητα, στη χρήση ενέργειας ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτώ λοιπόν τι, θεωρεί, συνέπειες θεωρείτε ότι θα έχει το σύστημα του backloading ή το να μην κάνουμε τίποτα αντίστροφα στις επιχειρήσεις. Η ΣΕΦΙ και οι άλλες μεγάλες επιχειρήσεις που εσείς εκπροσωπείτε και που έχουν κάνει σημαντική προσπάθεια ήδη. Αυτοί που θέλουν να λάβουν κάποια πρωτοβουλία για το κλίμα, τι συνέπειε θα δουν να τους πλήττουν. Ή μήπως τελικά βρεθούν με ένα μάτσο χαρτιά εκπομπών στα χέρια τους. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, ολοκληρώθηκαν εδώ οι ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χέρμαν για να απαντήσει. Βλέπετε ότι τα δύο τρίτα των προβληματισμών των βουλευτών είναι τα σχετικά με το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης, CDM. Είχαμε την, ο, στη συνεδρίαση εκείνη που το είχαμε συζητήσει πολλά θέματα να αντιμετωπίσουμε. Είχαμε εντοπίσει κάποια προβλήματα, τώρα βλέπουμε ότι αναδύονται και άλλα. Κύριε Μπότσεκ, εσείς εκπροσωπείτε επιχειρήσεις έντασης ενέργειας. Πρέπει να πω ότι το green economy σαν όρος, πράσινη οικονομία, εμένα δεν μου αρέσει. Δεν ε, τον δέχομαι, όπως δεν δέχομαι και τον όρο ε, θεά βιομηχανία εάν θέλω να προχωρήσω μια αναδιάρθρωση της παραγωγής και της ε, κοινωνίας, δεν νομίζω ότι θα πρέπει κάθε επιχείρηση να εγκαθίσταται σε έναν ε, πύργο από ατσάλι ή από μπετόν. Υπάρχουν διαφορετικές λύσεις. Επίσης, για την ε, λεγόμενη διαρροή άνθρακα, carbon leakage. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ μια επιχείρηση που μου είπε ότι κινδυνεύει από το carbon leakage ε, ακόμα και εταιρεία τηλεπικοινωνιών λόγω ακριβώς της, ή τουλάχιστον μία σημαντική με την ε, λύση που προτείνεται. Ενώ θα έπρεπε πιστεύουμε να εξαιρεθούν. Εδώ λοιπόν έχουμε περιλάβει όλες τις επιχειρήσεις ενώ εκείνοι οι οποίοι έχουν το καλύτερο την καλύτερη νομική υπηρεσία ή τους καλύτερους νομικούς συμβούλους μπορούν να καταφέρουν να εξαιρεθούν από τις διατάξεις και τα μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο ε, αυστηροί ή όχι. Θα πρέπει να δούμε τελικά ότι εκείνοι που κινδυνεύουν από το carbon leakage θα πρέπει να έχουν τη ε, διαφορετική μεταχείριση και τις άδειες. Όταν στο σύστημα εντάσσονται και επιχειρήσεις οι οποίες δεν κινδυνεύουν από το carbon leakage, ίσως τελικά στρεβλώνεται το σύστημα. Και θα ήθελα να μου πούν όλοι εδώ παρόντες πώς κρίνουν το σύστημα και τι προβλέπουν να φέρει η ενδεχόμενη αδράνεια, το να μην αναλάβουμε δράση δηλαδή και να μην εισαχθεί κάποια αλλαγή στο σύστημα. Εν τέλει, για τον κύριο Φόριστερ ε, που αναφέρθηκε στο χρυσού κανόνα, πιστεύω ότι αν πρόκειται να γίνει μια παρέμβαση στο σύστημα, θα πρέπει αυτή να είναι διατυπωμένη κατά τρόπο ώστε να δηλώνει ξεκάθαρα πως πρόκειται και μια εφάπαξ επέμβαση, έτσι ώστε όπως είπε και ο κύριος Βότσεκ, οι επιχειρήσεις, αλλά εν γέννη οι πάντες να έχουν στη θέση τους ένα σύστημα σταθερό, μέσο, αλλά καλύτερα ακόμη και μάκρο πρόθεσμα, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορούν να λειτουργούν, να παράγουν και να είναι αποδοτικό μέσα στην Ευρώπη. Γιατί θέλω να συνεχίσουμε να έχουμε και βαριά βιομηχανία στην Ευρώπη, βιομηχανία προ των υλών, εξωτερική βιομηχανία, ε, βιομηχανία χαλκού και το καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία μπορούμε να παράγουμε στην Ευρώπη θέλουν να παραμείνουν στην παραγωγή στην Ευρώπη, να μην χρειάζεται να τα φέρνουμε απ' έξω και από τα άλλα μέρη του κόσμου και βέβαια θα είναι κρίσιμη σημασία ε, η εξέλιξη ως προς τις εκπομπές, ως προς ανταλλαγές. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα τις απαντήσεις. Θα παρακαλέσω την κυρία Μπρι να λάβω το λόγο, παρακαλώντας όμως όλους τους ομιλητές να είναι σύντομοι, διότι έχουμε μέχρι τις 6.30 στη διάθεσή μας μόνο για να συζητήσουμε, γι' αυτό θα παρακαλώ ο καθένας να περιοριστεί στα 4 λεπτά για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με το ερώτημα για την ε, ε για τα χιτήρια και την χημική βιομηχανία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μειώσουμε το κόστος μας και να μειώσουμε τις εκπομπές μας. Αλλά επίσης η διαδικασία ε, συγκράτησης και αποθήκευσης άνθρακα είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλω να τονίσω ότι το ETS είναι η καλύτερη προσέγγιση χαμηλού κόστους και ο καλύτερος τρόπος για να μειώσει η βιομηχανία τις εκπομπές τους. Όλα εξαρτώνται από το αν θέλουμε να θέσουμε ένα τίμημα για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος ή όχι. Τώρα δεν μπορώ να προβλέψω βέβαια τις πελλοντικές ε, τιμές. Υπάρχουν πολλά άρθρα που λένε άλλα ότι θα υπάρξει ή μια προσωρινή αύξηση, μια προσωρινή μείωση και αυτό θα εξαρτάται από την μορφή του backloading. Αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρξει δράση άμεση για να δοθεί το απαραίτητο πολιτικό μήνυμα και να υποστηριχθεί η αξιοπιστία του συστήματος και μετά φυσικά μπορούμε να εξετάσουμε πιο μακροπρόθεσμα μέτρα. Τι θα γίνει αν δεν κάνουμε τίποτα τώρα. Είναι δύσκολο να προβλέπει κανείς, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό θα οδηγούσε σε προβλήματα με την αξιοπιστία του συστήματος. Είμαστε σε οικονομικές συνδίκες που δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει το 2008 και γι' αυτό χρειάζεται τάση. Ευχαριστώ κύριε Μπόσοκ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματα και εγώ εντυπωσιάζομαι από το επίπεδο κατανόησης και βαθιάς γνώσης της Επιτροπής σας για τα ζητήματα που συζητούμε εδώ πέρα. Και εγώ δεν υποστηρίζω την ε, ιδέα αυτή της πράσινης οικονομίας που θα οδηγήσει σε διάκριση μεταξύ διαφορετικών τομέων και διαφορετικών προϊόντων που παράγονται από τη βιομηχανία. Ακόμα και αυτοί που πιστεύουν σε κάποια μορφή πράσινης οικονομίας θα πρέπει να κατανοήσουν ότι όλα αυτά πρέπει να βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, σε πραγματική, στην πραγματική οικονομία, η οποία θα πρέπει να κληθεί να οικοδομήσει την πράσινη οικονομία. Πρέπει να έχουμε λοιπόν όλους αυτούς τους παραγωγικούς τομείς και να επιτύχουμε τη βελτίωση της ε, αποδοτικότητάς τους. Στον bus Eichhout πράγματι υπάρχουν εταιρείε που έχουν αποθέματα πιστοποιητικών και ίσως είναι έτσι ασφαλής για το άμεσο γιατί έχουν αυτά τα αποθέματα. Αλλά συγχρόνως υπάρχουν άλλες εταιρείε οι οποίες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τα χρήματα από αυτά που πήρανε στο παρελθόν σε δωρεάν πιστοποιητικά, διότι είχαν να αντιμετωπίσουν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Δεν είναι ότι ο τομέας Α ή ο τομέας Β έχει ένα μαξιλάρι από θεμάτων και μπορεί να κάτσει και να μην κάνει τίποτα. Κάτσει στα αυγά του και να μην κάνει τίποτα. Πιστεύω ότι αυτό μπορείτε να το ρωτήσετε και σε άλλους, σε τράπεζες, σε hedge funds, σε κερδοσκόπους. Τι κάνετε με τα πιστοποιητικά τα οποία έχετε στα χέρια σας. Αν τα έχετε κρατήσει ή αν τα έχετε ρευστοποιήσει. Αυτό είναι μια απόφαση που παίρνει κάθε εταιρεία. Έχουμε ακούσει να υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν μια ενιαία απάντηση σε αυτό το ερώτημα και ούτε υπάρχει μια ενιαία απάντηση στο ερώτημα του ποια είναι η τιμή του άνθρακα η οποία θα παροτρύνει την συγκράτηση και αποθήκευση άνθρακα. Αυτό το οποίο για μένα είναι σίγουρο είναι ότι η παρέμβαση που προτείνεται από την Κομισιόν και η οποία θα τύχει μάλλον απόψε μεγαλύτερης διευκρίνησης σημαίνει μια αύξηση κόστους για την ευρωπαϊκή οικονομία και για τα νοικοκυριά. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο πρέπει να θέσουμε ως υπεύθυνοι εμπλεκόμενοι είναι αν αυτό είναι το σωστό μήνυμα το οποίο θέλουμε να δοθεί και ιδίως σε μια κατάσταση όπου τουλάχιστον προς το παρόν η Ευρώπη είναι ο μόνος χώρος σε παγκόσμιο επίπεδο που έχει μια τιμή για τον άνθρακα αντίθετα με άλλους μεγάλους ανταγωνιστές μας. Για το ερώτημα. Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός σε σχέση με το κόστος δρόμος για να επιτύχουμε τους στόχους τους 2020 ε, Εγώ νομίζω ότι είναι σαφές ότι πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι. Τι άλλο θέλετε, υψηλότερε τιμέ ε, άνθρακα, αλλά σε ποιου τομεί. Δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να καθοριστούν οι τιμέ. Εμεί θα πρέπει να καθορίσουμε του στόχου και μετά να ακολουθήσουμε την οδό χαμηλότερου κόστου για την επιτεύξη των στόχων. Υπάρχουν νέε ριζικέ τεχνολογίε όπω και στη χαρτοβιομηχανία και στη χημική βιομηχανία θα θέλαμε να εφαρμοστούν αυτές τις τεχνολογίες. Πολλές από αυτές τις τεχνολογίες για να αναπτυχθούν χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις. Όπως και η έρευνα και η ανάπτυξη, όλα αυτά απαιτούν μια μεγάλη πολιτική πρωτοβουλία. Αλλά δεν είναι το ETS το σύστημα αυτό το οποίο θα δημιουργήσει τα απαραίτητα κονδύλια για κάτι τέτοιο σε βάρος της οικονομίας, της γενικότερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα σταματούσε εδώ. Ευχαριστώ. Για τον κατάλογο για την ε, λεγόμενη διαρροή άνθρακα. Ναι, φυσικά θα αναθεωρηθεί, ε, αν θυμάμαι καλά, το 2015. Είναι εν ε, εξελίξη αυτή η εργασία, η Κομισιόν εξετάζει όλες αυτές τις παραμέτρους, αλλά δεν έχει πολύ νόημα να πούμε ότι ο κατάλογος αυτός βασιζόταν στα 35 ευρώ και τώρα είναι στα 8 ευρώ ο τόνος του άνθρακα. Βρισκόμαστε σε μια βαθιά οικονομική ε, κρίση και δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει αμνούς με ερήφια. Το 2008 δεν είχαμε προβλέψει μια τόσο βαθιά ύφεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φόρεστερ. να σταθώ στο ερώτημα του Chris Davis. Σχετικά με τις συνέπειες της εφαρμογής του συστήματος. Οι συνέπειες, αν δεν υπάρξει το backloading, έχουμε συγκεκριμένες προσδοκίες. Ε, οι προσδοκίες αυτές της αγοράς λέγουν ότι κάτι πρέπει να γίνει, το θέμα είναι πόσο. Αν δεν συμβεί τίποτα τότε οι τιμές θα πέσουν περισσότερο γιατί ακριβώς οι προσδοκίες αυτές έχουν καθορίσει εν μέρη τις τιμές. Αυτή είναι μια άποψή μου βέβαια προσωπική και δεν εκφράζω μια επίσημη θέση της οργάνωσής μου. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι και με τη ρύθμιση του backloading οι περισσότεροι στην αγορά όπως είπε και η εκπρόσωπος της Επιτροπής σαν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί σε μία πραγματικά θα έλεγα πιεσμένη ή μάλλον σε αγορά, σε ύφεση, τότε δεν θα προσπαθήσει κανείς να κάνει τις επενδύσεις τις οποίες θα έκανε υπό πραγματικά καλύτερες συνθήκες. Το θέμα είναι το μακροπρόθεσμο, τι θα γίνει, εκεί είναι τα διαφορετικά τα μέτρα, αυτό έχουν, αυτά έχουν σημασία, τα υπόλοιπα δεν είναι σημαντικές αλλαγές. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία θα πρέπει να εξηγήσουμε στον φορολογούμενο σχετικά με το τι θα γίνουν με τα χρήματα αυτά έτσι ώστε να υπάρξουν καλύτερες επιδόσεις και σε επίπεδο γενικότερα οικονομικό. Ένα άλλο θέμα, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο δεν θα ήθελα να αγνοήσουμε είναι ότι αυτό το οποίο επίσης θα μπορούσε να χαθεί και είναι και αυτό μία από τις συνέπειες, είναι η αξιοπιστία της Ευρώπης και η αξιοπιστία του συστήματος περί του οποίου συζητάμε εδώ. Νομίζω ότι ακόμα και με τα προβλήματα που παρουσιάζει το σύστημα αυτό είναι ένα πραγματικά ζηλευτό σύστημα και αν χάσει αυτή την λάμψη θα έλεγα αυτό θα είναι αρνητικό για όλους. Ένα τελευταίο σημείο είναι ο λεγόμενος χρυσούς κανόν. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τους εμπλεκόμενους στην αγορά να κατανοήσουν ότι εάν μία ρύθμιση για το backloading ξεκινήσει, αυτό θα είναι κάτι το σπάνιο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση και εφόσον ακόμα και οι διαφορετικές ρυθμίσεις θα είναι σπάνιες ρυθμίσεις, είναι ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται γιατί ξέρουμε ότι δεν θα γίνονται συχνά. Μια διευκρίνηση μπορώ να ζητήσω. Ο Φόριστερ είπε ότι αν δεν υπάρξει το backloading τότε οι τιμές σαν κατάλαβα θα κατέβουν ακόμα περισσότερο. Αν υπάρξει το backloading πιστεύετε να αυξηθούν σημαντικά οι τιμές. Κοιτάξτε, όχι δεν θα αυξηθούν σημαντικά, γιατί όπως είπα οι σημαντικές αλλαγές στις τιμές εξαρτώνται, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση εν πάση περιπτώσει. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει την αγορά είναι οι διορθωτικές αλλαγές οι οποίες θα αφορούν το μέλλον και αυτές θα επηρεάσουν ε, τις τιμές. Κύριος Χέρμαν. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσαμε με, την, ε, με ένα απλό μοντέλο στην ε, μελέτη μας και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αν δεν γίνει τίποτα θα φτάσουμε στα 7 ευρώ, ενώ με ένα backloading ε, με 1,4 δις άδειε θα φτάσουμε σε μια τιμή 10 ευρώ για, τον, για την άδεια, το οποίο δείχνει ότι ακόμη και με μια με ένα πάγωμα, ε, ένα set aside που θα έχουμε ενδεχομένω, πάλι θα φτάσουμε στις ίδιες τιμές ε, μέχρι το 2020. Μιλάμε λοιπόν για συνέπειε. Ε, με το backloading μόνο ενός ή δύο ευρώ διαφοράς. Ακούστηκε ότι μπορεί οι κυβερνήσει να επιδιώκουν να εξασφαλίσουν νέα έσοδα με τις ε, προτάσεις αυτές για το ETS. Δεν θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό όμως, άρα δεν βλέπω πώς μπορούν να επηρεάσουν τις ε, τιμές για τις άδειε. Και ως προς τα διαρθρωτικά μέτρα, τι με διαρθρωτικά μέτρα θα πρότεινα εγώ. Με έναν μακροπρόθεσμο γραμμικό παράγοντα μείωσης μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημαντικό ποσοστό α, μείωσης του άνθρακα μέχρι το 2050. Πρόταση δική μου θα ήταν συνδυασμός του παγώματος του set aside και του, της γραμμικής ευθυσμίωσης. Για να φτάσουμε μέχρι τους στόχους του 2020-2030 θα πρέπει να πιέσουμε κάπως ε, τα αριθμητικά μας. Ε, δεν θα δώσω αριθμητικά στοιχεία συγκεκριμένα τώρα, αλλά νομίζω ότι αυτή θα ήταν η σωστή κατεύθυνση. Οι χώρες που έχουν ε, πρόβλημα προς τι χαμηλές τιμέ στι άδειε. Ε, κοιτάξτε, στη Γερμανία έχουμε μεγάλες ε, μονάδες φυσικού αερίου που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αντίστοιχε εγκαταστάσεις με βάση τον άνθρακα καινούριε εγκαταστάσει, καινούριε μονάδες φυσικού αερίου, που δεν μπορούν να ανταγωστούν παλιότερε παλιά τεχνολογία και αποτελεσματικότητας 30-35% μονάδες. Και αυτό όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και στην Αυστρία και σε άλλες χώρες. Άρα δεν είναι πολύ καλή κατάσταση. Για το CDM. Μέλλον δεν βλέπω. Ο κίνδυνος που διαβλέπω όμως είναι ότι θα επιδιώξουμε ένα υψηλότερο ποσοστό μείωσης και θα προσπαθήσουμε πάλι να καλύψουμε το κενό με ένα ε, μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης. Γι' αυτό θα προτιμούσα να μην δώσουμε μεγάλες ποσότητες CDM ως διορθωτικά μέτρα στις αγορές. Ευχαριστώ. Θα δώσω και το λόγο στον κύριο Μπέκη τώρα για να απαντήσει σε ερωτήσεις που τον αφορούν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ήθελα να απαντήσω στον ισχυρισμό της κυρίας Κόρχολα που λέει ότι η Κομισιόν είναι ο κυριότερος εχθρός του ETS. Είναι γεγονός ότι η πολιτική μας για την αποτελεσματικότητα της ενέργειας και την ε, προ... πρόοδο προς τα... τις ανανεώσιμες ενέργειες οδηγούν σε μείωση των εκπομπών. Εμείς είχαμε ένα πακέτο για τις ανανεώσιμες ενέργειες και τη μείωση των εκπομπών ταυτόχρονα και είχαμε προσαρμόσει τα μεν στα δε. Στην πρότασή μας για ενεργειακή απόδοση επίσης κάναμε σαφές ότι έπρεπε και πάλι να αναπροσαρμοστούν μεταξύ τους τα τρία αυτά στοιχεία. Αυτό ελέγχθηκε κατά τη διαπραγματεύσεις από την Κομισιόν. Ξέρουμε ότι αυτές οι πολιτικές πρέπει να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά οι στόχοι μας θα πρέπει να είναι συναρμόσιμοι μεταξύ τους και γι' αυτό θεωρούμε ότι το ETS πρέπει να αποτελέσει ένα κύριο πυλώνα σε όλα αυτά. Ένα δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι για τον απότερο στόχο του ETS. <clears throat> για μας ο τελικός στόχος είναι να δώσει ένα κίνητρο για επενδύσει σε οικονομία χαμηλού άνθρακα, χαμηλής χρήσης άνθρακα και καινοτομία αυτού του είδους. Δεν είναι θέμα κόστους, είναι υπέρ των επενδύσεων στις κατάλληλες τεχνολογίες του μέλλοντος. Και το τελικό μου σχόλιο είναι το εξής Επιβεβαίων αυτό που είπε ο κύριος Φόρεστε για τον χρυσού κανόνα. Όπως το βλέπουμε εμείς, οι παρεμβάσεις αυτές είναι εξαιρετικού χαρακτήρα. Είναι σπάνιες παρεμβάσεις. Δεν έχουμε σχέδια να τις επαναλάβουμε στο μέλλον και όπως έχετε δει, η Κομισιόν καθυστέρησε πολύ για να ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Μας υποχρέωσαν οι εμπλεκόμενοι να πάρουμε μια θέση για τα θέματα αυτά όταν οι τιμές εξακολουθούν να είναι τόσο χαμηλές κάτω από τα 10 ευρώ, θεωρούμε ότι είμαστε πράγματι στα πλαίσια μιας έκτακτης κατάστασης και ιδίως αυτά που ελέγχθηκαν για τους σταθμούς ενέργειας που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και που δεν είναι πια κερδοφόροι σε σχέση με τους παλαιάς τεχνολογίες σταθμούς ενέργειας με άνθρακα. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσιολογική και την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την πλούσια συζήτηση και θα καταγράψουμε όλα αυτά τα σχόλια και θα τα χρησιμοποιήσουμε στις συζητήσεις μας για την επόμενη φάση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέκερ. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να δούμε τι θα μας δώσει η Κομισιόν ε, και κύριε Μπόσαρκ, θέλω να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε στο ερώτημα του κυρίου Κριστέβης. Σας ευχαριστώ για το ε, ερώτημα αυτό για τα αυτοκίνητα, για τον στόλο αυτοκινήτου κατά κάποιο τρόπο. Το 2008 διατυπώθηκε αυτή η οδηγία και ξέρετε ότι υπήρχε η επιμονή ορισμένων σημαντικών εμπλεκομένων στο ETS να επομείνουν να υπάρχει εκ των προτέρων μια κατανομή πιστοποιητικών, δηλαδή μια αυτοκίνητο βιομηχανία να πάρει αποφάσεις για τα επόμενα 10 χρόνια σε σχέση με τον αριθμό των αυτοκινήτων που θα παρήγαγαν. Αυτό είναι ακριβώς κάτι για το οποίο ο Γιώστεν Μπέικερ είχε επιμείνει. Τώρα, όταν δεν έχουν αγοραστεί τα αυτοκίνητα, έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο τα διαφορετικά μέτρα τα οποία προτείνετε εσείς θα πρέπει να ληφθούν μετά το 2020. Να σκεφτούμε για μια πιο δυναμικού χαρακτήρα κατανομή, λαμβάνοντας υπόψη την βιομηχανική παραγωγή, την οικονομία εν γέννη και όλα αυτά που συμβαίνουν στο περιραίον περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ και ο Χριστέβης. Ευχαριστώ. Ε, ο Σώσα Βάγνερ έχει τώρα το λόγο για να κλείσει. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να παρατηρήσουμε είναι η ποιότητα και η ποσότητα των απόψεων τις οποίες εξέφρασαν και οι ευρωβουλευτές και οι εμπειρογνώμονες που πήραν μέρος σε αυτή τη συνάντηση. Πάρα πολύ σύντομα γιατί δεν έχουμε πλέον χρόνο να έχουμε προβλήματα θα έλεγα ουσίας και έχουμε και προβλήματα διαδικασικά. Αυτό φάνηκε από όλες τις παρεμβάσεις και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα προβλήματα ουσίας θα έλεγα αποτελούν μια σειρά θεμάτων τα οποία θα πρέπει να βασιστούμε σχετικά με την οδηγία, επί τη βάση μάλλον της οδηγίας για την αποδοτικότητα της ενέργειας την οποία εγκρίναμε σχετικά πρόφατα. Πάνω εκεί θα πρέπει να βασιστούμε. Και μετά υπάρχουν και διαδικαστικά θέματα. Αυτά τα διαδικαστικά, κατ' και σε επίπεδο γενικών αρχών είναι ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τον ρόλο συναπόφασης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως επίσης ε, και τον σημαντικό ρόλο της πολιτικής στον τομέα ε, του περιβάλλοντος που θα πρέπει να ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι βέβαιος ότι η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σίγουρα θα βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση για τα προβλήματα στα οποία αναφερθήκατε. Ευχαριστώ κύριε Σούζο Βάγνα. Και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ θερμά όλους όσοι έλαβαν μέρος στη συζήτησή μας σήμερα, όλους τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν μέχρι τις Βρυξέλλες για να μας μιλήσουν, την Επιτροπή, τον κύριο Ντεβέκη, την Επίτροπο βεβαίω και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ γιατί μας προσφέρατε τη δυνατότητα να εργαστούμε πολύ εντατικά επί τρεις ώρες για το θέμα των ανταλλαγών εκπομπών. Το σύστημα ETS, όπως είπα και από την αρχή, είναι το ισχυρότερο μέσο ε, ανά τον κόσμο για τις ανταλλαγές εκπομπών. Εγώ προσωπικώς αισθάνομαι υπερήφανο προσωπικά που έχουμε επιτύχει να εγκαθιδρύσουμε ένα τέτοιο σύστημα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να μιλάμε με πιο πατριωτικούς τόνους, να ενστερνιστούμε δηλαδή το σύστημα αυτό και να λέμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, πώς αλλιώς μπορούμε να το προαγάγουμε. Και ταυτόχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε να μην τα ε, παραγνωρίζουμε, αλλά να προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις ουσιαστικές και μακροπρόθεσμες. Περί αυτό πρόκειται. Και αυτό σημειώνω από τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν σήμερα για το backloading ότι είναι μια συγκεκριμένη εφάπαξ επέμβαση, όπως πρέπει και να είναι, που ίσως θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε για την τέταρτη περίοδο, εάν είναι χρήσιμο να αντιδρούμε, να αντιδράσουμε δεδομένων των σημαντικών πιέσεων της συγκυρίας για να βρούμε τι είδου μέσα μπορούμε να βρούμε για αντίδραση. Για το Συμβούλιο ETS βεβαίως εάν και άλλοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό θα πρέπει να γίνει η συζήτηση και να ληφθούν οι αποφάσεις του τι είδου ε, φόρουμ θα ε, αποφασίζει ένα συμβούλιο ETS, παραδείγματι, για την ε, ένταξη νέων μελών, αλλά και τους λοιπούς όρους. Πάντως, ευχαριστώ πολύ. Συζητούμε μια πρόταση, η οποία μόνο χρόνο μας εξασφαλίζει, μας κερδίζει λίγο χρόνο και πρέπει να διευκρινίσουμε βεβαίως πώς θα το επιτύχουμε αυτό. Από το χέρι μας περνάει πιστεύω ότι με τρόπο παραγωγικό, στραμμένη προς το μέλλον και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προτάσεις, ιδέες, υποδείξεις που ακούστηκαν σήμερα όλες κυριολεκτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο το απόγευμα η ώρα 3, για τους συναδέλφους τώρα μιλάω, Κάνουμε την ακρόαση του υποψηφίου Υπουργού για θέματα δημόσιας υγείας. Καλό σας βράδυ και όσοι μένετε έξω από τις Βρυξέλλες, καλή επάνωδο.